Πολύ καλημέρα σας. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, θα ξεκινήσουμε το σημείο 2 που είναι ανακοινώσεις ε, του Προέδρου για τις αποφάσεις που έλαβαν χθες οι συντονιστές. Και μετά, επαναλαμβάνω, θα ψηφίσουμε. Το Πρόεδρο χθε λοιπόν έλαβε ορισμένε αποφάσει σε σχέση με τι ε, γνωμοδοτήσει. Προσθέθηκαν στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χέλμερ, από το EFD. Μετά, ε, δεύτερη έκθεση, μάλλον γνωμοδότηση για τα επιβατικά οχήματα το ΕΛΚ. Και τρίτη, για την γνωστή γνωμοδότηση για την μία και μόνη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ECR θα αναλάμβανε αυτή τη γνωμοδότηση. Βέβαια, είπαμε ότι θα περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι συνάδελφοί μας από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, την ΑΦΚΟ, και μετά θα αναλάβουν οι συνάδελφοι της ομάδας CCR την γνωμοδότηση. Πρώτα λοιπόν οι συντονιστές αποφάσισαν να περιμένουμε την απόφαση της ΑΦΚΟ και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Επίσης, Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε η επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γαλλικίας από τις 12 έως 13 Φεβρουαρίου. Δεν υπήρξαν ενστάσεις σε ό,τι αφορά την πρόταση του κυρίου Μπουλόν που θα είναι και ο επικεφαλής, ο αρχηγός της αντιπροσωπείας αυτής, ο οποίος ζήτησε να πάει μια μέρα νωρίτερα η αποστολή για λιμένες υποχρεώσεις που είχε ο ίδιος. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στη Γαλλικία, υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων για τα διάφορα σημεία του προγράμματος και αποφασίστηκε οι συμμετέχοντες στο στην αποστολή και λέγοντας αυτό εννοούμε τα επίσημα μέλη και επιτόπιοι βουλευτές, οι βουλευτές. Είπαμε ότι θα περιμένουμε ε, να δούμε και πώς θα έχει ολοκληρωθεί τελικά το πρόβλημα. Κυρία Μιράντα, βλέπω ότι είναι εδώ. Θα ζητήσουμε τον κύριο Μπουλόν που θα είναι ο αρχηγός της ε, αντιπροσωπείας αυτής να καθορίσει μια ημερομηνία για να συναντηθούν ε, όλα τα μέλη αυτής της αποστολής. Επίσης αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος του συναδέλφου και φίλου Μποστινάρου να συναντηθούμε και με τον δήμαρχο της πόλης του Βίγκο. Και υπόθηκε επίσης ότι καλό θα ήταν να συναντηθούμε όχι μόνο με τον δήμαρχο του Βίγκο, αλλά και με όλους τους ε, ε, δημάρχους ε, των, της ευρύτερης περιοχής του Δέλτα του Βίγκο. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να συναντηθούμε με όλους αυτούς τους δημάρχους. Κυρία Όκερ, μα δεν νομίζω ότι λάβαμε κάποια απόφαση είπαμε θα δούμε τους αναφέροντες και τις αρχές, αλλά ε, δεν αποφασίσαμε ακριβώς ποιους θα συναντήσουμε. Είπαμε θα το δούμε στην επόμενη συνέντευξη των συντονιστών, νομίζω. Μα θα έχουμε επιστρέψει από τη Γαλλικία και μετά θα γίνει η επόμενη συνέντευξη των συντονιστών. Άρα η αποστολή αυτή θα πρέπει να αποφασίσουμε. Νομίζω ότι αυτό είπαμε ε, στη συνεδρία των συντονιστών. Είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Βίγου και άλλου δημάρχου, αν βέβαια στο επιτρέπει το πρόγραμμά του και είναι διαθέσιμη. Η αποστολή όμω είναι αυτή η οποία θα λάβει την απόφαση. Κυρία Όκεν. Εγώ φοβάμαι μην απογοητεύσουμε του αναφέροντε. Γιατί δεν με ικανοποιήσει και πολύ τρόπο με τον οποίο τα συζητήσαμε χθε. Πρόεδρος, ωραία, σας ευχαριστώ Μάργαρετ για τις διευκρινήσεις αυτές. Λοιπόν, έπειτα έχουμε το επόμενο σημείο μια ακόμη επίσκεψη στην ε, Ισπανία σε σχέση με τις αναφορές που σχετίζονται με τον νόμο για τις ακτές, λέει Κώστας. Θα αποφασιστεί το πρόγραμμα σε μια επόμενη συνεδρία, θα τα δουν και η ομάδα εργασίας τα σχετικά. Και ένα τρίτο σημείο ήταν μια επίσκεψη στην Ελλάδα σε σχέση με τα απόβλητα και απορρίμματα και άλλα θέματα. Ο κ. Σαλαβράκος που δεν είναι σήμερα εδώ ζήτησε αν είναι δυνατόν να αλλάξουν ημερομηνίε γιατί δεν θα μπορούσε να είναι τότε, αλλά όπως είπε η Γραμματεία δεν έχουμε πολλές δυνατότητε. Προβλέπεται λοιπόν αυτή η επίσκεψη για τα τέλη Μαΐου στην Ελλάδα, επίσκεψη στην Ελλάδα. Επίσης, η ομάδα Άλντε, φιλελεύθερη δηλαδή, και συγκεκριμένα η κυρία Μπέρμαν, είπε χθε στι συνεδρίες των συντονιστών ότι υπάρχει στη Δανία ένα πρόβλημα για τις υιοθεσίες παιδιών. Ζήτησε η κυρία Βέρτμα να το δούμε πολύ γρήγορα, γιατί είναι ένα σοβαρό ζήτημα. περισσότεροι συντονιστές συμφώνησαν και αποφασίσαμε το συντομότερο δυνατό να διεκπαιρεώσουμε αυτό το θέμα. Ένα άλλο ζήτημα είναι το αίτημα της ομάδας του ΕΛΚ. Και συγκεκριμένα ο κύριος Μπολά, ο οποίος ενδιαφέρεται να συζητηθούν αναφορές που έχουν να κάνουν με την ε, Γαλλία και συγκεκριμένα είναι ένα πρόβλημα με ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην Άντι, στην περιοχή Notre Dame de Έχουμε όμως ορίσει ποιε θα είναι οι μας για το έτος αυτό. Άρα καταρχήν δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε μια ακόμη επίσκεψη. Όμως, τελικά τι θα γίνει. Θα συζητηθεί στην Επιτροπή Αναφορών για το Μάρτιο ή τον Απρίλιο Ανάλογα με το τι θέματα έχουμε να συζητήσουμε στη μερική διάταξη, επαναλαμβάνω το θέμα θα τεθεί είτε το Μάρτιο είτε τον Απρίλιο στην Επιτροπή μας. Εγκρίθηκε επίση η μερική διάταξη για μια κρόαση για την ημέρα των πολιτών. Στις 19 συγκεκριμένα. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην για διάταξη, ενώ τη χθεσινή συνεδρία των συντονιστών. Ο κύριο Γιάρο όμω μου λέει ο Ντέβιντ Λό ότι θέλει να μιλήσει. Θέλει να πει κάτι Πέτερ. 19 είπατε. Ποιο μήνα όμω, κύριε Πρόεδρε. Α, ναι, με συγχωρείτε, το ξέχασα ο Πρόεδρο. 19 Φεβρουαρίου. 19 Φεβρουαρίου. Το θέμα αυτό λοιπόν για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο να απευθύνει έκκληση στην διάσκεψη των Προέδρων, διότι έχουμε το πρόβλημα με τις διερευνητικές αποστολές και το χρονοδιάγραμμα, το πότε θα γίνουν. Έχουμε και την πράσινη εβδομάδα. Και έχουμε θέμα χρόνου. Δεν μπορούμε να κάνουμε δύο ταξίδια παράλληλα. Οι διαβεντικές αποστολές έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα καταρχάς και Δεύτερον, μπορούμε να περιορίσουμε σε μία ή δύο μέρες τις διερευνητικές αποστολές, να το συζητήσουμε αυτό, το πώς θα το κάνουμε, πώς θα κάνουμε τις ε, διερευνητικές αποστολές, να, να μας προταθεί μία ημερομηνία, να δούμε ποιος θέλει να πάει. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και των ε, υπολείπων αποστολών και αντιπροσωπιών. Ε, έχουμε δύσκολο πρόβλημα γενικότερα και αλλά δεν μπορούμε να εξισώνουμε τις ερευνητικέ αποστολές με τις άλλες αποστολές ε, και αντιπροσωπείες. Πρέπει να δούμε να μην υπάρχει σύγκρουση στο πρόγραμμα. Γι' αυτό σας ε, καλώ να παρέμβετε. Uh, uh, Μάργαρετ, πρώτα απ' όλα. Πάρα πολύ σύντομα. Θα είμαι σύντομη. Συμφωνώ με τον Πιτεγιάρ. Πιστεύω πως ε, πρέπει να απευθυνθούμε όχι μόνο στον πρόεδρο, αλλά και στους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Είναι μια απόφαση που θα τη λάβει διάσκεψη των προέδρων και βλέπετε ότι αυτό επαναλαμβάνεται και λόγω των πράσινων εβδομάδων πρέπει να επαναπρογραμματίσουμε τις ερευνητικέ αποστολές. Μετά υπάρχουν προβλήματα στο πρόγραμμα των άλλων αντιπροσωπιών. Αυτό ε, ιδιαίτερα τον Οκτώβρη θα είναι μεγάλο πρόβλημα. και πρέπει να απευθυνθούμε και στους Προέδρους και στους Γενικούς Γραμματείς ταυτόχρονα και να τους πούμε ότι θέλουμε περισσότερη ευελιξία και περισσότερες δυνατότητες. Κυρία Μπέρμαν, ε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ το υποστηρίζω αυτό πλήρως. Μπορείτε να καταλάβετε όλοι πώς ε, μπλοκάρουμε τις εργασίες μας και όπως υπόθηκε αυτές οι διερευνητικές αποστολές στην Επιτροπή Αναφορών είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με, αυτό που κάνουμε στις άλλες επιτροπές. Ωραία. Ακούστε, ακούστε. Σημειώσαμε, σημειώσαμε τις παρεμβάσεις σας, αυτά που είπατε. Σημειώνουμε λοιπόν αυτά που θίξατε, τα τρία αυτά σημεία. Όμως στην τρία των συντονιστών θα μπορούσαμε στην ημερήσια διάταξη να γράψουμε το σημείο αυτό. Άλλωστε και οι τρει που λάβετε το λόγο είστε συντονιστέ, άρα μπορούμε να τα δούμε στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Και όπως λέει ο Ντέβιτ, θα μιλήσουμε και με, τους, ε, με τις αρχές, ο πρόεδρος, για αυτό το θέμα. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή τίποτα σχετικό με τη σύνδεση των συντονιστών, θα περάσουμε στο σημείο 13. Έχω ένα πρόβλημα. Έχουμε την... Έχω εδώ την ημερησία διάταξη στα Ιταλικά. Παρακαλώ, δώστε μου αυτή στα Ισπανικά. Ξέρω γιατί μου έδωσαν την ημερησία στα Ιταλικά, την νόμιζα θα είναι η κυρία Ματσόνη, αλλά δεν μπορεί η κυρία Ματσόνη. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, David. Έχουμε λοιπόν την έκθεση επί της ειδικής έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την έρευνα σχετικά με την προσφυγή 2591-2010 κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επέκταση αεροδρομίου της Βιέννης. Κυρία Όκεν, έχει στήσει το λόγο. Μου είπαν οι διερμηνείς ότι θα ήταν ε, καλύτερο, πιο ευγενικό να μιλήσω τη γλώσσα μου, τα δανέζικα. Θα το προσπαθήσω λοιπόν. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους πολύ για την εξαιρετική συνεργασία. Μάλιστα, γελούν με, το... με τη διερμηνία, δεν ξέρουν αν είναι στο σωστό κανάλι οι συνάδελφοι. Είχαμε λοιπόν εξαιρετική συνεργασία. Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα. Τώρα έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκέλος των ε, συμβιβασμών και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλά. Να πω ότι θέλαμε να έχουμε μία σωστή νομική βάση στο τελευταίο στάδιο της ψηφοφορίας. Και το λέω αυτό διότι πολύ συχνά βλέπουμε ότι όταν η νομοθεσία δεν είναι αρκετά αυστηρή, πολλές φορές το αδύναμο μέρος κινδυνεύει. Ο πολίτης, το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως εμείς είμαστε ως αντιπρόσωποι των πολιτών υπεύθυνοι σε αυτή την Επιτροπή ειδικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ, ιδιαίτερα τους Αυστριακούς συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάργκριτ. Äh, Θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο, κατά εξαίρεση. Καταρχάς, ε, να πω ότι το οι δεν είναι κάτι αυτονόητο, εκτός από την εισηγήτρια η οποία ε, ηγήθηκε με εξαιρετικά δημιουργικό τρόπο της ε, έκθεσης αυτής και οι σκιώδεις εισηγητές εξίσου αξίζουν συγχαρητήρια και οι συντονιστές και οι πολιτικές ομάδες, διότι όλοι είχαν πνεύμα συνεργασίας. Και αυτό ήταν προφανέστατο από τότε που άρχισε ο Ευρωπαίος Δημοσιολευτής να ασχολείται με το θέμα. Και επίσης, να μην ξεχάσουμε και την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εισήλθε σε ανοιχτό διάλογο. Ήταν υποδειγματική η συνεργασία Εργαστήκαμε καλά πάνω σε ένα αρκετά προβληματικό θέμα προς ε, το συμφέρον των πολιτών. Κοιτάξαμε πώς θα τους αντιπροσωπεύσουμε καλύτερα. Κοιτάξαμε τις συνέπειες, ιδιαίτερα με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και να πω και ότι η επικοινωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη αξιολογήθηκε πολύ θετικά και μπορούμε και στο μέλλον να αναμένουμε ε, τέτοια θετικά στοιχεία συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπέκερ. Μετά από το μουσικό Ιντερλούδιο, μπορούμε να περάσουμε στον κύριο Μποστινάρου και κάποιο άλλο θέλει το λόγο. Λοιπόν, γρήγορα παρακαλώ γιατί έχουμε πολλά σημεία στην Ταξί, Κύριε Μποστινάρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο η μουσική μας σταματά τελικά. Πραγματικά, καταφέραμε να συντάξουμε μια εξαιρετικά εντυπωσιακή έκθεση και να ευχαριστήσω τη Μάργαρετ και τον κύριο Μπέκερ και όλους τους συναδέλφους και πραγματικά ο τρόπος που συντάχθηκε η έκθεση αυτή ήταν υποδειγματικός και καταφέραμε να έρθουμε σε συμβιβασμό και αυτό είναι εντυπωσιακό, ιδιαίτερα διότι το θέμα είναι τόσο ευαίσθητο, ιδιαίτερα διότι το νομικό πλαίσιο ήταν λίγο πολύ ασαφές Ωστόσο, η Επιτροπή μας κατάφερε να προτείνει νέους κανόνες, τους οποίους έλαβε υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τους λαμβάνει υπόψη από εδώ και στο εξή. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τους αναφερόμενους και ως το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Και τέλος ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό, διότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι όσοι συμμετείχαν και και συνεισεφεράν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εξυπηρετήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες. Ήταν ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα και για την αξιοπιστία της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Μάργαρετ. Κύριε Μπέργμαν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ και για τη μουσική υπόκρουση και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλες τις πλευρές, διότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο συνέχεια. Έχουμε κάτι... Είχαμε κάτι δύσκολο, αλλά εξαιτία της επικοδομητικής συνεργασίας καταφέραμε να βρούμε μία λύση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.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 ο πρόεδρος. Υπέρ λοιπόν συμβαστικής κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, α, μία ψήφος κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η εννέα και αυτή είναι συμβιβαστική με την 11. Όχι. Εννέα συμβαστική λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά δύο ψηφικατά. κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές κατά. Λοιπόν, η επόμενη είναι κατά τμήματα. Στην παράγραφο 13. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ψήφι υπέρ. Λοιπόν, μου ζητείτε επαλήθευση για το τμήμα 2. Λοιπόν, εσκόντε καλά τα χέρια σας. Στην παράγραφο 13 λοιπόν το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Δεύτερο με Μάργαρετ. Μάργαρετ. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα της παραγράφου 13. Ποιοι είναι υπέρ, έτσι. Λοιπόν, Πριν είπε κατά ο πρόεδρος, τώρα λέει υπέρ. Λοιπόν, ποιοι είναι κατά τώρα. Ποιοι είναι κατά τώρα. Okay. Τελικά τι γίνεται. Απορρίπτεται τελικά. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Λοιπόν, απορρίπτεται. 10 προς 7 ήταν η αναλογία των ψήφων. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα, λοιπόν, και περνάμε τώρα στην τροπολογία 12. Καταπίπτει, λέει ο γραμματέας. Λέει εδώ στα χαρτιά μας ότι αν εγκριθεί συμβιβαστική καταπίπτη, λέει ο κ. Πουστινόρ έχει δίκιο, μου φαίνεται. Τι έγινε όμως εδώ πέρα. Πράγματι μπορεί να καταπέσει γιατί τα στοιχεία περιλάμβανε, περιλαμβάνονταν συμβιβαστική. Μπορούμε να πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Λοιπόν, οκ, συμφωνούμε κατά 12, περνάμε στην 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. 13, 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στο recital 1. Την τολική σκέψη 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ της έκθεσης. Ε, μετράτε, εντάξει, ωραία. Κατά, αποχές, συγχαρητήρια, ομόφωνα υπέρ, 19 ψήφι υπέρ. Υπάρχει και μία αποχή βέβαια, αλλά δεν υπάρχει καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια λοιπόν κυρία Άουκεν. Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε τώρα λοιπόν στο σημείο 14 και θα δώσω τη σκητάλη της Προεδρίας στην κυρία Παλιαδέλη. Good morning to all of you. Καλημέρα σε όλους. γνωμοδότηση για την εκτίμηση περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων σε τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με εισηγητή τον κύριο Χουντή. Κύριε Χουντή, θα θέλετε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. που να επικρατήσει τάξη θα πω διάφορα εθιμοτυπικά. Θέλω να σας καλημερίσω όλους και όλες. Θέλω να καλημερίσω και τους διερμηνείς. Το θέμα που συζητάμε είναι σοβαρό. Πρόκειται για την τροποποίηση της οδηγίας 2011 του 92 και που αφορά στις εκτιμήσεις των επιπτώσεων από έργα δημόσια και ιδιωτικά στο περιβάλλον. Όταν ένα θέμα είναι σοβαρό στην Ελλάδα, λέμε πως σηκώνει καφέ, χρειάζεται καφέ. Ελπίζω να έχετε πει ένα πρώτο καφέ. Εύχομαι να έρθει καφές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκτός αν τα μέτρα λιτότητας έκοψαν και τον καφέ στις συνεδριάσεις. για εσάς κύριε Όχι δεν, ε, καταλάβατε το λέω να ησυχάσει λίγο η αίθουσα αλλά έχει και τη σημασία του για να συγκεντρωθεί η προσοχή μας στο θέμα που μας αφορά. Μπαίνω λοιπόν, μπαίνω λοιπόν στο θέμα επαναλαμβάνοντας ότι είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα είναι και σημαντική η δική μας γνωμοδότηση που συλλογικά θα διαμορφώσουμε για ένα θέμα, για μια πολιτική που είναι βασικό εργαλείο για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι τι επιπτώσεις υπάρχουν από τα δημόσια και ιδιωτικά έργα στο περιβάλλον. Υπάρχει αυτή η οδηγία, πάνω από 20 χρόνια εφαρμόζεται έχει ενσωματωθεί στις εθνικές ένομες τάξεις, αλλά, αλλά υπάρχουν ανησυχίες ως προς την εφαρμογή της. Αυτό μπορεί να το έχει ο καθένας μας ως εμπειρία από τη χώρα του, αλλά θέλω να σας πω ότι στην Επιτροπή μας, δηλαδή στην Επιτροπή Αναφορών, έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλές αναφορές, πάρα πολλές αναφορές από τους πολίτες της Ευρώπης από όλα σχεδόν τα κράτη όπως μελετήσαμε με τους συνεργάτες ότι υπάρχουν πρακτικές που καταστρατηγούν την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Πιο αναλυτικά, κατά την καταγραφή και τη στατιστική που έγινε και την αίσθηση που έχουμε και οι ανησυχίες εκφράζονται στο γεγονός ότι τα προβλήματα όσο αφορά την εφαρμογή ή γενικά την υλοποίηση μιας τέτοιας οδηγίας, πέρα από τη γενικά ελλειπή εφαρμογή, έχουν σχέση με ότι υπάρχουν έργα στα οποία δεν είναι υποχρεωτική η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει σε κράτος ή και εργολάβους, γιατί μιλάμε για δημόσια και ιδιωτικά έργα, να την αποφεύγουν. Υπάρχει μια τυπολατρία στην ύπαρξη, όταν προκύπτει τέτοιο θέμα, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία όμως δεν στέκεται στην ουσία του περιεχομένου. Υπάρχουν προβλήματα όσο αφορά την ενημέρωση των ενδιαφορεμένων. Τα χρονικά περιθώρια στη διαβούλευση δεν είναι τέτοια που να μπορέσει να γίνει ουσιαστική ε, ε, διαβούλευση και να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή στην καταγραφή των επιπτώσεων και τι θα γίνει. Και βεβαίως υπάρχει και η πρακτική, θα ήθελα να το προσέξετε αυτό, σαλαμοποίησης των έργων σε μικρότερα, ώστε να μην απαιτείται η, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έτσι να περνάει χωρίς αυτό την απαραίτητη πολιτική άσκηση πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος. Θέλω να σας ενδιαφέρω αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, έστω καθυστερώντας λιγάκι, ότι οι περισσότερες αναφορές που έχουν έρθει στην Επιτροπή μας όλα αυτά τα χρόνια αφορούν αρνητικές επιπτώσεις <clears throat> και σε μεσαία και μεγάλα έργα υποδομής. Αναφέρεται τα θέματα σχεδίων για τις γέφυρες στην περιοχή Λουάρ κοντά στην Ορλεάνη. Επίσης αναφέρονται σε απειλές κατά μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, παραδείγματος χάρη στην Ιρλανδία, ο αυτοκινητόδρομος που διασχίζει και καταστρέφει την περιοχή του μνημείου Τάρα και επίσης έχουμε αρκετές αναφορές από πολίτες της Ιταλίας, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας για θέματα χωροθέτησης και κατασκευής αποβλήτων. Επανέρχομαι λοιπόν στην πρόταση που κάνει η Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις. Αυτά τα προβλήματα, αγαπητοί συνάδελφοι, τα κωδικοποιεί σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις, σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα είναι πρώτον διαδικασίες ελέγχου, η δεύτερη είναι η ποιότητα και η ανάλυση της ε, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η τρίτη κατηγορία, η τρίτη ομάδα προβλημάτων ελλείψεων που διαπιστώνει και η ίδια Επιτροπή γι' αυτό προβαίνει στην πρόταση για την τροποποίηση αυτής της οδηγίας, αφορούν τους κινδύνους ανακολουθιών ε, και τη σχέση που έχει η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με άλλα νομοθετήματα και προτείνει ορισμένες τροποποίησεις. Για να μην σας κουράζω, είναι η πρώτη άλλωστε συζήτηση που κάνουμε σήμερα, υπάρχει ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα που το έχετε υπόψη σας, αναφέρεται στο πρόγραμμα, πότε θα ξανακουβεντιάσουμε δεύτερη φορά τρίτη φορά, θα γίνουν τροπολογίες, θα ξαναψηφίσουμε και επομένως για τις ανάγκες της πρώτης παρουσίας και της πρώτης συζήτησης θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένες από τις, τροποποίησει τροποποίησεις που προτείνονται θέτοντας και κάποια ερωτήματα. Ερωτήματα προς την Επιτροπή που θα μας αποσαφηνίσουν καλύτερα τι σκέφτεται και τι προτίθεται να κάνει. Νομίζω ότι είναι εκπρόσωπος εδώ της Επιτροπής και τον παρακαλώ στη σειρά του το Προεδρείο θα κανονίσει να μα δώσει αν μπορεί σήμερα κάποιε διευκρινήσεις στα θέματα που θα αναφέρω παρακάτω. Υπάρχει στο άρθρο 1 και στην παράγραφο 3. Εδώ λίγο για να το συνδεθείτε με το θέμα υπάρχει στην τροποποίηση, την υφιστάμενη τροποποίηση εξαίρεση στις μελέτες εκεί περιβαλλοντικών επιτόσων όταν πρόκειται για λόγους εθνικής άμυνας. Αυτό έχουμε μέχρι τα τώρα. Τώρα με την προτινόμενη τροποποίηση από την πλευρά της ε, Επιτροπής προστίθεται σε αυτές τις εξαιρέσεις και τα θέματα κατάστασης έκτακτης ανάγκης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Εδώ τίθεται ερώτημα, γίνεται και κριτική. Κάτω από το όνομα ή κάτω από την κατηγορία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ε, επιτρέψτε μου να το πω έτσι γιατί, μπορεί να γίνουν σημεία και τέρατα. Η επίκληση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας μπορεί να διευρύνει τον κατάλογο των εξαιρέσεων και να έχουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές στο, περιβάλλον από τα έργα αυτά για τα οποία αναφερόμαστε. Επίσης, στην ίδια, στο ίδιο άρθρο και στο άρθρο 4, όπως καταλαβαίνετε καθορίζει τις κατηγορίες όπου χρειάζεται η Επιτροπή που υπάρχει εξαίρεση, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα και θα έλεγα επίκαιρη όσο αφορά φαινόμενο των καιρών, προστίκη για την οποία έχω ισχυρότατε ενστάσει, θα το κουβεντιάσουμε. Λέει λοιπόν ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για έργα που εγκρίνονται με ειδική νομοθετική πράξη. Εδώ κατά τη γνώμη μου ανοίγει παράθυρο μεγάλο για την καταστρατήγηση της οδηγίας. Επιτρέψτε μου αγαπητοί συνάδελφοι να σας μεταφέρω <clears throat> την εμπειρία την ελληνική. Μέσα στις συνθήκες της κρίσης και του μνημονίου έχουμε το νόμο 4014 του 2011 που χαρακτηρίζεται από τη λογική να επιταχύνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης από την άποψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατόπιν τούτου ελαστικοποιούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις στο όνομα να γίνουν κάποια έργα διότι υπάρχει ανάγκη, διότι υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ λοιπόν επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου αυτό το σημείο τι σημαίνει η ειδική εθνική νομοθετική πράξη, σας ανέφερα το παράδειγμα. Στο άρθρο 2 στέκομαι στα πιο βασικά όπως σας είπα ε, και στην παράγραφο 3 η πρόταση της Επιτροπής ορίζει, ζητάει, απαιτεί να διαμορφωθεί μια αρχή αρμόδια για να διευκολύνει τη διαδικασία χορήγησης άδεια για κάθε έργο. Εδώ ακριβώς είναι το ερώτημα προς την Επιτροπή. Τι ακριβώς εννοεί. Τι είναι αυτή η Επιτροπή. Ποια θα είναι η σχέση της με τις ήδη υφιστάμενες αρμόδιες εθνικές αρχές θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Θα είναι υπεράνω όλων των άλλων των σημερινών υφισταμένων η νέα αρμόδια επιτροπή που προτείνει η Επιτροπή. Θα ήθελα να διευκρινιστεί αυτό το θέμα και επίσης στο ίδιο άρθρο, αναφέρομαι στο άρθρο 2, ε, περιλαμβάνει τη συνέργεια, τη σχέση της οδηγίας ΕΠΕ ε, επιπτώσεων περιβαλλοντικών, ε, μάλλον ε, ερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μαζί με άλλα, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μαζί με άλλα περιβαλλοντικά νομοθετήματα. Κατά τη γνώμη μου είναι θετικό αυτό, είναι θετικό, αρκεί να μην <laughs> κρύβεται μια απόπειρα να μειωθούν οι ασφαλιστικές δικλίδες. Στο άρθρο 3, για να συντομεύω, ε, οι τροποποίησεις που προτείνεται είναι να προσαρμοστεί η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα νέα φαινόμενα που έχουμε ή μάλλον σε, προβλήματα όπως, ε, σε θέματα όπως βιοπικιλότητας και κλιματικών αλλαγών. Εδώ όμως υπάρχει κάτι που πάλι μας δημιουργεί, μου δημιουργεί ερωτήματα και που νομίζω ότι η αοριστία αφήνει παράθυρο και εδώ. Ε, αναφέρομαι στην, προσθήκη συγγνώμη, τις λέξεις σημαντικές όσο αφορά τις άμεσες και έμεσες επιπτώσεις ενός έργου. Και η λέξη σημαντικές δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Επομένως τι εννοούμε και ποιες θα χαρακτηρίζονται σημαντικές ούτως ώστε να έχουμε αυτή την επισήμανση. Τα άρθρο 4 και 5 υπάρχει ένα θέμα, το έχουμε δει στην Επιτροπή Αναφορών, ότι υπάρχει ε, πρόβλημα και έλλειψη συνοχής στον τρόπο που τα κράτη διεξάγουν, κάνουν τους ελέγχους. Σε πολλές φορές η, αυτός ο έλεγχος επαφίεται σε εθνικές αρμόδιες επιτροπές. Ωστόσο, ε, ε για να τεκμηριωθούν αυτές οι πληροφορίες, για να τεκμηριωθεί όλο αυτό το πράγμα. Η εκτίμηση που έχει έρθει πολλές φορές, επαναλαμβάνω, στην Επιτροπή Αναφορών, ότι αυτές οι μελέτες, αυτή η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πολλές φορές στερείται αντικειμενικότητας. Διότι η μελέτη, η ευθύνη αυτής της, μάλλον η ευθύνη αυτής της μελέτης ανατίθεται στον κύριο του έργου. Δηλαδή δεν κρίνει αντικειμενικά αν πράγματι υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Επομένως, επειδή είναι κρίσιμη σημασίας, θα ήταν καλό αυτή τη ε, μελέτη να την έκανε, να γινόταν ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος, όχι ο κύριος του έργου. Ε, και για να μην σας κουράζω τελευταία παράγραφος, αναφέρομαι πάλι ξαναλέω στις σημαντικές τροποποίησεις, είναι <clears throat> το θέμα που τίθεται στο άρθρο 8, στην παράγραφο 2, όπου αναφέρεται ότι η αρμόδια επιτροπή, αρχή μπορεί ουσιαστικά να χορηγεί άδειες ακόμα και για έργα με σοβαρέ αρνητικέ επιπτώσει στο περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση, αν έχει σοβαρέ επιπτώσει, πρέπει να απορρίπτεται. Ή να υπάρχει δυνατότητα α, για, για πρόσθετα μέτρα που να περιορίζουν αυτές τις ζημιές. Και επομένως εδώ χρειάζεται προσοχή τι σημαίνει αυτό και πώς γίνεται όταν πρόκειται περί οφθαλμοφανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Θα έλεγα καταρχήν να απορρίπτεται. Αν υπάρχουν εναλλακτικέ προτάσει πρέπει να αναφέρονται και δεύτερο πώς αποκαθίστανται οι ζημιές και ποιος τις πληρώνει αυτές τις ζημιές από ήδη ε, ας το πούμε διαπιστωμένες αρνητικές επιπτώσεις ε, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Ε, αυτά θα ήθελα να πω για να μην σας κουράζω περισσότερο. Ε, ξαναλέω ότι υπάρχει ένα θέμα ποιος μηχανισμός κάνει αυτή τη μελέτη και ποιος παρεβαίνει διορθωτικά, ποιος επιβαρύνεται το κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα λίγο πριν περιμένω την απάντηση της Επιτροπής ε, και τελειώνω υπογραμμίζοντας ε, χωρίς χαριτολόγημα πια ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Ελπίζω να, από την πρώτη παρουσίαση να σας έπεισα γι' αυτό και περιμένω τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ανοχή Εγώ ευχαριστώ κύριε Κουντή. Μας πείσατε ως ένα βαθμό, αλλά περιμένω να ακούσουμε τις απόψεις του κυρίου Αμπατζή από την Επιτροπή. Ο κύριος Αμπατζής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χουντή. Θα, συνήθως στην Κομιτέτη Πετησιών μιλάω στα ελληνικά, αλλά λόγω του θέματος αυτού που αφορά όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλα τα κράτη-μέλη θα μιλήσω στα ε, αγγλικά. So, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα σχόλια. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι η αναθεώρηση ακολουθεί την έκθεση για το αεροδρόμιο της Βιέννης όπου τονίστηκε ότι ως Επιτροπή αναμένουμε την ε, αναθεώρηση και τη γνωμοδότησή σας, διότι όπως θα δείτε και με την εκτίμηση επιπτώσεων, ένα από τα κύρια θέματα που ήταν η αφορμή της πρότασής μας, ήταν η εφαρμογή της οδηγίας μέσω συγκεκριμένων ε, παραπώνων και αναφορών. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που ο κύριος Χουντής έθιξε και ανέφερε αυτές τις ανησυχίες σχετικά με τα προβλήματα ε, εφαρμογής αυτής της οδηγίας που εφαρμόζεται εδώ και πάνω από 27 χρόνια. Θα ήθελα να αναφέρω δύο γενικά σχόλια ε, ως προστήκη στα όσα είπε ο κύριος Χουντής και μετά να απαντήσω στους διάφορους προβληματισμούς που έθιξε για τα συγκεκριμένα άρθρα. Καταρχάς, ο γενικός στόχος της ε, αναθεώρησης ήταν η διόρθωση των ε, εντοπισμένων προβλημάτων εφαρμογής, αλλά και να γίνει στοχασμός πάνω στις ε, προκλήσεις, τις περιβαλλοντικές ε, και κοινωνικές και είμαι σίγουρος ότι η οδηγία αυτή εναρμονίζεται με τον υπάρχοντα κανονισμό. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το, τις αποφάσεις και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο μας έχει δώσει αρκετή εμπειρία και πολλά διδάγματα και προηγούμενο για το πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες περιπτώσεις. Ε, επίσης, υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι αυτής της οδηγίας. Ο πρώτος στόχος είναι η εισαγωγή ή η ενίσχυση των στοιχείων που έχουν σχέση με την ποιότητα των εκθέσεων ΕΠΕ, αλλά και όλης της διαδικασίας ΕΠΕ γενικότερα. Το δεύτερο στοιχείο ήταν να ενισχυθεί η πολιτική συνοχή, αλλά και να διασφαλιστεί εφαρμόζεται με απλοποιημένες διαδικασίες. Τώρα, όσον αφορά τα σχόλια του κυρίου Χουντή σχετικά με τα άρθρα, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τα παραρτήματα της οδηγίας, ιδιαίτερα τα παραρτήματα 3 και 4, στα οποία έχουμε πολλές τροπολογίες, ουσιαστικές τροπολογίες, τις οποίες θα θα εφαρμόζουμε μαζί με τις ε, διατάξεις. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 1.3, υπήρχε μία εξαίρεση στην οδηγία για κάποια έργα τα οποία εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Τώρα προσθέσαμε και έργα όχι μόνο για πολιτική προστασία, αλλά έργα τα οποία είναι απάντηση σε ανάγκες, σε πολιτικές ανάγκες. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και πολλές φορές δεν υπάρχει χρόνος για ε, ΕΠΕ και αυτό μας έχει δείξει και η εμπειρία. Έτσι λοιπόν το προσθέσαμε μαζί με τις ε, περιπτώσεις πολιτικ... Ε, πολιτικής ανάγκης και τις περιπτώσεις πολιτικής άμυνας. Επίσης έχουμε ενισχύσει την διατύπωση πριν από αυτό, λέγοντας ότι, αυτό, ότι αυτά τα έργα θα πρέπει να εξαιρούνται εάν εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς και έργα εθνικής άμυνας ή έργα που απαντούν σε περιπτώσεις ε, πολιτικής έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, ας πούμε, και μαζί με αυτό θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα πάρκινγκ. Θα γίνει εξαίρεση μόνο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο ή και στο πάρκινγκ του. Το σκεπτικό λοιπόν ήταν να εξαιρέσουμε συγκεκριμένα και αποκλειστικά έργα που έχουν να κάνουν με εθνική άμυνα ή απάντηση σε, περι... Ε, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτή η εξαίρεση προσθέθηκε βασισμένη στην ε, εμπειρία που έχουμε με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίση, στο άρθρο 2, παράγραφος 4, υπάρχει μία εξαίρεση που δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και η οποία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ε, έχουν εξαιρέσει την οδηγία σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει. Και η εμπειρία μα από το 1985 μέχρι τώρα έχει δείξει ότι η απάντηση σε περιπτώσει έκτακτη ανάγκη είναι μια εξαίρεση σε αυτό το άρθρο. Και αυτό θέλαμε να το λάβουμε υπόψη και να το προσθέσουμε στι συγκεκριμένε εξαιρέσει. Θα θέλαμε όμω να διασφαλίσουμε την Επιτροπή σα ότι έχουμε λάβει υπόψη όλους τους προβληματισμούς και θα φροντίσουμε ώστε να μην γίνεται κατάχρηση αυτής της εξαίρεσης. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο τώρα, η δυνατότητα των κρατών μελών να εξαιρέσουν ένα έργο το οποίο εξαιρείται μέσω νομοθετικής πράξης, υπήρχε ήδη στην οδηγία. Υπάρχει εκτεταμένη νομολογία και πρόσφατες υποθέσεις, για υπόθεση Μπόξους για παράδειγμα, και η νομολογία αυτή διασφαλίζει τις ε, προϋποθέσεις εφαρμογής. Και αυτό που κάναμε εμείς στην Επιτροπή ήταν να προσθέσουμε μία υποχρέωση αναφοράς για τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται αυτή η διάταξη. Και μέσω αυτού θέλουμε να ελέγξουμε πώς χρησιμοποιούν τα κρατημέλη την εξαίρεση αυτή, αλλά να πω ότι η εξαίρεση μέσω νομοθετικών πράξεων είναι σπάνια. Χρησιμοποιείται σπανιότατα ορισμένα κρατημέλη όπως η Δανία, η Ιταλία, το Βέλγιο ή η Ελλάδα τη χρησιμοποιούν αν όμως αισθάνεστε ότι πρέπει να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις εξαίρεσης, τότε να το δούμε. Αυτό ίσως είναι αναγκαίο. Τώρα, όσον αφορά το σημείο του άρθρου 2, παράγραφος 3, αν κατάλαβα καλά, έχετε κάποιες ανησυχίες με την τελευταία πρόταση για τον ε, διορισμό αρμόδιας αρχής που θα διευκολύνει τη διαδικασία έχετε θετική άποψη σχετικά με τις ε, υποχρεώσεις ε, ύπαρξης ενός συντονιστή στην όλη διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διάταξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, παράδειγμα, φανταστείτε ότι έχετε ένα, ένα χώρο καύσης απορριμμάτων που είναι κοντά σε ένα χώρο, σε μια περιοχή Natura 2000. Χρειάζεστε ΕΠΕ, άδεια, σύμφωνα με την οδηγία βιομηχανικών εκπομπών. Φανταστείτε λοιπόν ότι και για την αρμοδιαρχή και για εκείνον που διεκπεραιώνει το έργο, η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοφόρος. Με αυτή λοιπόν την οδηγία και με την ε, εισαγωγή αυτής της υποχρέωσης αναφοράς θέλουμε να εξομαλύνουμε τη διαδικασία και να διασφαλίσουμε περισσότερη συνοχή ανάμεσα στις ε, πολιτικές. Το σκεπτικό όμως δεν ήταν τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν καινούργιε αρμόδιες αρχές. Όχι, το σκεπτικό είναι να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να συγκεντρώσουν όλες τις σχετικές αρμόδιες αρχές και να τις υποχρεώσουν να συνεργασούν έτσι ώστε να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν ομαλότερα. Ήταν δύσκολο, όπω καταλαβαίνετε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ποια αρχή είναι αρμόδια. Ήταν θέμα επικουρικότητα. Το θέμα ήταν, ε, και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, ήταν να συγκεντρώσουμε όλε τι αρμόδιε αρχέ σε ένα τραπέζι και να του αναγκάσουμε να συνεργαστούν. Και προ όφελο του περιβάλλοντο και προ όφελο του ίδιου του έργου που θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 3. Ε, χαίρομαι που αναγνωρίσατε την ανάγκη εξυγχρονισμού των ΕΠΕ και να ληφθούν υπόψη η κλιματική αλλαγή και η οδηγία για το κλίμα ή για τη βιοπικιλότητα ή για κινδύνους καταστροφών. Ισχύει ότι στο άρθρο 3 δεν υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες. Ήταν πιο γενικό. Όλα αυτά τα ζητήματα όμως ε, αναφέρονται εκτενέστερα στα παραρτήματα και στην οδηγία προσπα... Θύσαμε να είμαστε πιο σύντομοι και στα παράρτηματα να επεξηγήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά και, να αναφερθούμε στη βιοποικιλότητα, για παράδειγμα. Αυτά τα θέματα δεν θα επηρεάσουν όλα τα project. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε ιδιαίτερα το διοικητικό φορτό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, οι ανησυχίε καταστροφή σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο που βρίσκεται δίπλα από μια φάρμα. Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος καταστροφής είναι μεγαλύτερος από ό,τι σε άλλες. Τέλος, για την προσθήκη της λέξης significant, σημαντικό στο άρθρο 3. Προσθέσαμε αυτή τη λέξη, το significant, βρίσκεται παντού στην οδηγία και στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στο οποίο είναι και ο κύριος στόχος. Η ΕΠΕ έχει να κάνει με την αξιολόγηση σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γι' αυτό το θεωρήσαμε σημαντική βελτίωση και το προσθέσαμε στο άρθρο 3. Στα άρθρα 4 και 5 βλέπω ότι στα σχόλιά σας τα σχολιάσατε μαζί. Θα ήθελα να τα χωρίσω όμως και να πω ότι στο άρθρο 4 και σε συνδυασμό με το παράρτημα 3 προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, ιδιαίτερα με τα έργα στα οποία δεν απαιτείται ε, απαραίτητα ΕΠΕ και να ασχοληθούμε και με το ζήτημα της σαλαμοποίησης, το οποίο προκύπτει πολύ συχνά, και να θέσουμε ιδιαίτερα κριτήρια στο άρθρο 3 που να ασχολούνται με αυτό το θέμα και έτσι ελπίζουμε όχι να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να λύσεις όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον να δώσουμε τα μέσα στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό, ώστε να μπορέσουν να έχουν καλύτερο έλεγχο τη περίπτωση. Όσον αφορά το άρθρο 5, υπάρχει μια πολύ σημαντική διάταξη που έχει να κάνει με την ποιότητα τη οδηγία ΕΠΕ και ίσως αυτή είναι μία από τις κύριες διατάξεις της ε, οδηγίας και αυτό διαφάνηκε και από τα σχόλιά σας, διότι στο άρθρο 5 ασχολούμαστε με θέματα όπως τις ε, λογικές εναλλακτικές λύσεις, τι είδους πληροφορίες μπαίνουν σε μία έκθεση ΕΠΕ, πού πρέπει να εστιάσουν οι αρμόδιες αρχές και οι διεκπαιρεωτές. Και στο άρθρο 5 επίσης προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το, με ζήτημα της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της ε, πληροφορίας, ότι να δούμε τι χρησιμοποιούν, ποιο μοντέλο χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη, να δούμε τις εκθέσεις που καταρτίζονται από αρμόδιους και εμπειρογνώμονες στον κάθε τομέα. Επίσης, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, μαζί με το άρθρο 8 παράγραφος 4, αναφέρουμε ανησυχίες για την ισχύ, για την ημερομηνία. Για παράδειγμα, οι ΕΠΕ χρειάζονται πολύ καιρό για να καταρτιστούν. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε κάποιε ΕΠΕ οι οποίε έχουν καταρτιστεί 10 χρόνια πριν εγκριθεί ένα project. Αυτή είναι μια πολύ μακρά περίοδο. Το περιβάλλον μπορεί να έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν με αυτά τα άρθρα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Τελειώνω με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στο άρθρο αυτό, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, υπάρχει μια σημαντική διάταξη. Στην παράγραφο 1 προσπαθούμε να πούμε ποιες πληροφορίες πρέπει να μπαίνουν στις αποφάσεις, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο λήφθη υπόψη το περιβάλλον. Στην παράγραφο 2 ε, αναφέρονται προϋποθέσεις γιάτσι και αυτό θα επηρεάσει έργα τα οποία θα έχουν σημαντικά και αρνητικά και σημαντικέ και αρνητικέ επιπτώσεις. Να πω ότι το σκεπτικό και η φιλοσοφία της οδηγία δεν έχει αλλάξει. Πριν την αναθεώρηση αλλά και με την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής μπορούμε να εξακολουθήσουμε να εγκρίνουμε έργα που έχουν αρνητικέ επιπτώσει για το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, για παράδειγμα, ναι, μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε ένα ένα χώρο καύσης απορριμμάτων δίπλα στην Ακρόπολη, ας πούμε, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη εάν μπορεί να κατασκευαστεί ένα τέτοιο έργο που έχει αρνητικέ επιπτώσεις. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε την, τις πληροφορίες από πού προέκυψαν και να τις δούμε με όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο τρόπο και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προσθέτοντας μια υποχρέωση για τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την επίβλεψη και την εφαρμογή μέτρων αποζημίωσης, αποτελεσματικών μέτρων αποζημίωσης και προσπαθούμε να μην κάνουμε την ΕΠΕ απλά μία εκτίμηση σε χαρτί. Όχι, προσπαθούμε μέσω της οδηγίας να διασφαλίσουμε ότι αυτό που, έχει, που υπάρχει στο χαρτί θα εφαρμοστεί και στην πράξη. Σε γενικέ γραμμέ δεν έχει αλλάξει λοιπόν πάρα πολύ. Ελπίζω να σα ικανοποίησαν οι εξηγήσει μου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε προχωρούμε στις, Η κυρία Άουκιν ζήτησε το λόγο. Yeah, to... Uh, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον uh, κύριο Χουντή και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και θέλω να πω ότι πραγματικά περιμένουμε ανυπομονησία τη δουλειά που και εμείς θα εκπονήσουμε σε σχέση με την οδηγία αυτή. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε και επαρκή χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί εμείς εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά και πολύπλοκα ζητήματα. Για την Επιτροπή μας, αν όχι όλες, πάντως οι περισσότερες ε, αναφορές ασχολούνται, αφορούν την οδηγία αυτή που είναι μεν καλή, αλλά η εφαρμογή της το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ αυτό. Και είπαμε λοιπόν ότι περιμένουμε με απομονησία να ε, αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτήν. Κάποια σχόλια τώρα. Χαίρομαι που είπατε κι εσείς ότι είστε κατά της αλαμοποίησης. Γιατί πραγματικά μας εξοργίζει όταν βλέπουμε να γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Και έχουμε ακούσει και κάποια κριτική και του Δημοσιολαβητή για την Κομισιόν. Όταν μιλάτε για την επικουρικότητα δηλαδή, θα πρέπει να έχετε υπόψη ε, και το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Πρέπει να το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα πάρα πολύ σοβαρά και με τον ορθό τρόπο. Το είδαμε στην Αυστρία, για παράδειγμα. Χρησιμοποιήθηκε αυτό το επιχείρημα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια άλλη αρχή ε, για την εκτίμηση, την αξιολόγηση ε, του έργου. Μόνο ο ίδιος το αξιολογεί. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν αυτά που σας είπα υπόψη. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι εμένα τουλάχιστον θα με ανησυχούσε πάρα πολύ και το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Λαμβάνονται υπόψη, προστατεύεται τα δικαιώματα των πολιτών, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της οδηγίας ΕΠΕ είναι και η συμμετοχή των πολιτών. Θα πρέπει να τους ακούμε τους πολίτες και γνωρίζετε όπως και εγώ ότι έχουμε να κάνουμε με μεγάλους εργολάβους, με πάρα πολλά χρήματα και οι εργολάβοι χρησιμοποιούν και την επιρροή που τους δίνουν αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, εμείς ε, έχουμε καθήκον, έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πολιτών και να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με δίκαιο τρόπο και ειλικρινή. Σε ό,τι αφορά τώρα το κατεπήγον ή τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Οι Ιταλοί ε, το φωνάζουν πάντα, ούτε καν δηλαδή, αλλά τέλο πάντων. Πάντα ε, μιλάνε για επίγον, για κατάσταση έκτακτη ανάγκη ε, και έρχονται και οι φαντάροι, οι στρατιώτε, μπλοκάρονται τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε. Εντάξει, φυσικά και δεν μπορούμε να βάλουμε τη χωματερή στην Ακρόπολη δίπλα ή έναν αποτεφρωτή απορριμμάτων και κοντά. Εντάξει δεν αρκεί αυτό να το πούμε. Το θέμα είναι να δούμε ε, αν τηρείται και η δημοκρατία, γιατί κάθε χώρα θα αποφασίσει. Το θέμα είναι όμως να μην αφήνουμε παραθυράκια με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και δεν είναι μόνο η φύση, μιλάμε και για την πολιτιστική κληρονομιά που και αυτή μας ενδιαφέρει. Και πολλές φορές έχουμε δει φαινόμενα διάφορα. Βέβαια δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα εδώ. Πάντως ε, χάρηκα που είπατε ότι έχετε αντιληφθεί τα βασικά προβλήματα, όπως είπε και ο κύριος ε, Χουντής βέβαια και τα μας τα περιέγραψε. Καλό θα ήταν βέβαια και η Επιτροπή Ένβη ε, να επιληφθεί με τρόπο αποτελεσματικό για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η οδηγία και πρέπει να είναι και ως δυνατόν πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς αμφιβολία είναι μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση και οι αναφορές που έχουμε το δείχνουν και όλες ότι υπάρχουν ένα σώρο προβλήματα στον περιβαλλοντικό τομέα που έχουν σχέση με την οδηγία αυτή έπειτα. Από τη μία πρέπει όντως να έχουμε ε, διαβουλεύσεις, από την άλλη όχι και τόσο πολύ. Και να πω ότι θα έπρεπε να συναντηθούμε και οι συντονιστές ε, και οι σκιώδες εισηγητές και να εργαστούμε καλά και σοβαρά. Το πρόβλημα τώρα, ποιο είναι τα προβλήματα. Στην, ποιότητα των αναλύσεων, των ε, αξιολογήσεων και της ίδιας της διαδικασίας. Γιατί πολλές φορές βλέπω στις αναφορές που έχουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην ε, εναρμόνιση και έχουμε απόδειξη από τις αναφορές που λαμβάνουμε ότι αυτές οι ΕΠΕ είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Έπειτα χρειαζόμαστε ακριβώς αυτές ε, τις ΕΠΕ ουδετερότητα και αμεροληψία. Και τέλος, χρειαζόμαστε πιθανό, δυνατότητες τροποποίησης της διαδικασίας. Δηλαδή, όταν ας πούμε κάποιο project έχει ήδη διεκπαιρεωθεί, υπάρχει, τότε έχουμε πρόβλημα. Πώς θα το αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Και αυτό με απασχολεί. διότι οι αναφέροντες έχουν α πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει β πληροφορίες και μετά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν συνδυάζονται αυτές οι πληροφορίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν καλύτερο διάλογο για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας όσον αφορά τα επιμέρους άρθρα. Ένα, φυσικά και πρέπει να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε για τις εξαιρέσεις. Οι φυσικές καταστροφές είναι κάτι που μου έρχεται στο μυαλό. Στην περιοχή μου, όταν για παράδειγμα βρίσκονται άνθρωποι σε κίνδυνο επειδή έχει σπάσει ένα φράγμα και το νερό θα πλημμυρίσει μια περιοχή προστατευμένη, πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις. Επίσης, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τα στρατιωτικά έργα. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σχεδιάζει ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα ιδιωτικά έργα και στα κρατικά έργα. Πού θα υπάρχουν εξαιρέσεις, σε ποια από τα δύο. Πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση τα έργα και να, υπάρχει, να συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικές, οι σωστές ε, ΕΠΕ. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και να είμαστε σαφέστεροι. Άρθρο 2. Αυτή η αρχή των, ε, της συγκέντρωσης των αρμόδιων αρχών είναι κάτι που χαιρετίζω. Έχω και παραδείγματα και από την ε, Τσεχία, όπου εκεί πέρα υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές ε, για το περιβάλλον δεν είναι καλά ε, συνδεδεμένες, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, ο ένας πάει στον άλλο, στέλνεται ο ένας από τον άλλο στον καϊάφα κτλ. κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια, μια, ένα σημείο που συγκεντρώνονται όλα και συνεργάζονται. Τώρα, άρθρο 4, επίσης σημαντικό. Τα έργα που έχουν σχέση και με το πρασίνισμα, άρθρο 5, Λέξη κλειδί, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, φυσικά. Πρέπει να γίνει μια αμερόληπτη και αντικειμενική ΕΠΕ. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε εδώ να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της ΕΠΕ. Ποιος την παραγγέλνει, γιατί την παραγγέλνει. Άρθρο 8 τώρα. Εδώ θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα, να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να πούμε τι πληροφορίες χρειάζονται, πώς λειτουργεί η διαδικασία. Τι γίνεται με την επιτήρηση, με τον έλεγχο. Καταλαβαίνω βέβαια ότι το θέμα του ελέγχου είναι κάτι που αφορά την Επιτροπή και τα κρατημέλη και δεν είναι απόλυτα αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής. Αλλά να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι πρέπει και οι συντονιστέ και οι συντονιστέ να συζητήσουμε καλά και να δούμε από κοινού τι θέση θα λάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Ε, κύριε Μποστινάρου, παρακαλώ να είστε σύντομο γιατί. Ε, you have to be quick. Ναι, να είστε σύντομο παρακαλώ. It's very kind of you. Είναι πολύ ευγενέ που ζητάτε μόνο από μένα να είμαι ε, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα είμαι πειθαρχημένο, θα είμαι σύντομο. Λοιπόν, ναι, αυτό πρέπει να είναι το πιο σημαντικό σημείο ε, της ε, θητείας μας, της εντολής μας. Να απαντήσουμε δηλαδή ε, στα, στις ανησυχίες του Ευρωπαίου πολίτη. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Ε, έτσι ώστε το νέο νομικό ε, ε, νομοθετικό πλαίσιο που θα αποτελέσει βέβαια και το πεδίο εφαρμογής του νέου δημοσιονομικού πλαισίου να είναι ορθό. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είτε δεν έχουν ήδη απαντηθεί, είτε έχουν απαντηθεί αλλά με τρόπο ασαφή. Ας πούμε, πώς μπορεί κανείς να έχει ουδετεωρότητα, αμεροληψία, ε, αντικειμενικότητα σε αυτές τις μελέτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, το πάντα υποσυζήτηση, αν όχι υποαμφισβήτηση. Νομίζω ότι εμείς σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί έτσι ώστε να μην αφήσουμε καμία δυνατότητα συνενοχής ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ε, μια εταιρεία η οποία καλείται ε, να διενεργήσει την ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και τον ανάδοχο κτλ. Να μην υπάρχουν τέτοιου είδους συνάφειες ή συνενοχές. Δεύτερον, θα πρέπει να αποσαφινιστούν οι όροι ε, ε, ο, κατά τους ε, οποίους καθίσταται υποχρεωτική στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη. Τι μπορεί να αποφασιστεί, ποιος μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει μία SP γιατί από αυτό το σημείο απορρέουν πολλά προβλήματα. Θα πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή πότε είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αυτή ε, η στρατηγική μελέτη. Επίσης, αναφέρθηκε ήδη, θα πρέπει να αποσαφινιστούν οι όροι ε, με τους οποίους διοργανώνονται οι δημόσιες ακροάσεις, ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει το κοινό, συμμετέχουν οι πολίτες στις ε, ε, διαβουλεύσεις. Ξέρουμε ότι στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, και στην Ιταλία και αλλού, πολύ συχνά είναι φτιαχτές αυτές οι διαβουλεύσεις, είναι στημένες, πώς να σας το πω. Καλούν δηλαδή τους φίλους και τους φίλους των φίλων και κάνουμε μια φιλική κουβεντούλα και αυτό τελικά καθίσταται ε, και αποβαίνει μάλλον καταστροφικό. Αυτά είναι τα σημαντικά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Επίσης, ε, δεν ε, έχει αποσαφινιστεί το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα είτε των αναφερόντων είτε ε, των πολιτών γενικά. Για πολλά χρόνια τα κράτη-μέλη εκόφευαν κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να ξέρουν πότε είναι υποχρεωμένοι να ε, απαντήσει. Και η Κομισιόν θα πρέπει να ξέρει και θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς πότε είναι υποχρεωμένοι να απαντήσει ή να αντιδράσει. Γιατί το να αφήνουμε τα πάντα στις ελληνικές καλένδες δεν λύνει τίποτα αναβάλλεται, αναβάλλεται και τελικά χάνεται η υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, υπάρξει δεσμευτικό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί με την πάροδο του χρόνου, αφενός ξεχνιούνται πολλά πράγματα ή αφετέρου και πιο σημαντικό, μπορεί εντωμεταξύ να έχουν επιτελεστεί σημαντικότατες καταστροφές. στα μεγάλης κλίματος, κλίμακος ε, ε, ε, προγράμματα, πια, κυρίως αυτά που σχετίζονται με την ενέργεια, είτε είναι εξορρεκτικές διαδικασίες, είτε είναι ε, αγωγή, όπως το North Stream ή South Stream ή άλλοι. Όταν μιλάμε για θερμοελεκτρικούς σταθμούς ή τέτοιου είδους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ποια είναι η θεσμική απάντηση ή ποια είναι η θεσμική πίεση μετά από την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, εάν βεβαίως προβλήματα υφίστανται. γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτού του είδους τα προγράμματα μπορεί ε, να αναφέρονται ε, ε, εμπλεκόμενοι από διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται λοιπόν, πώς μπορούμε, δεν μπορεί η Βουλγαρία π.χ. μόνη της να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο ζήτημα όταν υπάρχουν εμπλεκόμενοι και πέραν των συνόρων. Τελική παρατήρηση θα ήταν ευτυχές, αλλά μάλλον αφελές, να θεωρούμε ότι ε, στο μέλλον ε, μπορεί να γίνονται πράγματα χειρότερα με, την, με τις ΕΠΕ. Γιατί εάν αρχίσουν να εφαρμόζονται προγράμματα χωρίς σε καμία ε, σοβαρή πρώτερη αξιολόγηση και μελέτη επιπτώσεων, αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στον τελικό μιλητή. Ε, πρέπει να πω το εξής. Ζήτησα να είστε ε, γρήγορος γιατί έχουμε εδώ ένα πρόβλημα με τη σλοβακική διαρμηνία. Θα πρέπει να πάμε αμέσως ε, μετά την ολοκλήρωση αυτή τη συζήτηση στο σημείο 22 διότι στις 10.30 ο Διερμηνέας από Σλοβακικά και προς φαντάζομαι θα πρέπει να φύγει. Γι' αυτό. Κύριε Μιράντα, αν μπορείτε γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση, κυρία Πρόεδρε, και γιατί αφορά, αναφέρεται στους πολίτες, αλλά και γιατί αφορά τον έλεγχο της εφαρμογής ε, της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Οι περισσότερες ανακοινώσεις ή καταγγελίες που λαμβάνω από πολίτες έχουν να κάνουν τη συγκεκριμένη οδηγία όλος περιέργος. Οι περισσότερες επαναλαμβάνω και αυτό γιατί δεν συμμετέχουν επαρκώς οι πολίτες, δεν ε, ζητείτε διαβούλευση μαζί τους και σας μιλάω με φράγματα, σας μιλάω για φράγματα, για χρυσορυχία, για ε, χιτά, ε, για το φράκινγκ, την υδρορογμάτωση και ούτω καθεξής. Και βέβαια κυρίως για την εφαρμογή του δικτύου Natura. Νομίζω λοιπόν ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση και η δυνατότητα να αποφύγουμε με πρόσχημα την κατάτμιση των έργων, να γίνεται η απόπειρα ε, παράκαμψης της κοινωτικής νομοθεσίας, αυτό μπορεί να μας δώσει μια μεγάλη δυνατότητα, ούτω ώστε τελικά να εφαρμόσουμε την κοινωτική νομοθεσία με αυστηρότητα ε, από πλευράς κρατών μελών. Και εκεί έγκυται μέχρι τώρα η αδυναμία, το πρόβλημα. Και αυτή η ιδέα τη συμμετοχή των πολιτών νομίζω ότι πρέπει να την ε, στηρίξουμε περισσότερο, γιατί δεν είναι. Είναι αρκετά αδύναμη στην πρόταση τη Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα υποβάλουμε σχετικά τροπολογίε στην ομάδα του κ. Χουντή. Ευχαριστώ. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούν να πούν δύο λόγια ο κ. Χουντή και ο κ. Αμπατζή ε, όσον αφορά το ζήτημα. Αλλά αν δεν θέλουν, αν, δεν έχετε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό να μας πείτε, να περάσουμε στο 22. Καλό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτη παρατήρηση, γιατί θα είμαι σύντομος, είναι γιατί πράγματι πρέπει να έχουμε χρόνο για να το συζητήσουμε. Και να συζητήσουμε και με τους συντονιστές. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να το αλλάξουμε το, το χρονοδιάγραμμα, και να μας δώσει περισσότερο χρόνο, το τελικό χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να το κουβεντιάσουμε φάνηκε από τη συζήτηση. Το δεύτερο που θέλω να σας πω ε, αγαπητοί συνάδελφοι και στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, από ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση, η, τα προβλήματα ή τα ερωτήματα, οι τροπολογίες που θα κατατεθούν και από μένα στο σώμα και στα παραρτήματα και από τους άλλους συναδέλφους, είναι δύο κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ανησυχίες για την ελλειπή εφαρμογή της σημερινής οδηγίας και πρέπει να ενισχυθεί ούτως ώστε να έχουμε λιγότερα περιθώρια. Και το δεύτερο που οφείλω να σας πω είναι η ανησυχία μου και φαντάζομαι και άλλων από τη λογική που αρχίζει να επικρατεί ως κατεύθυνση σε σχέση με την οικονομική, την κοινωνική κρίση ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη και αυτή η ανάπτυξη τουλάχιστον στη δική μου τη χώρα επιδιώκεται με διαδικασίες fast track επομένως που δεν παρακάμπτουν το περιβάλλον επομένως οι εξαιρέσεις, οι ευελιξίες κτλ είναι σίγουρο ότι θα αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η τρίτη Να σας πω ένα παράδειγμα πολύ σύντομα. Έκτακτη ανάγκη. Τι σημαίνει έκτακτη ανάγκη. Πάρτε ε, στη χώρα μου και αλλού. Χώρους εναπόθεσης ε, απορριμμάτων το πρόβλημα χρονίζων, χωματερές, φτάνει σε έκτακτη κατάσταση, δηλαδή κλείνουν τα χρονοδιαγράμματα, έρχονται τα πρόστιμα και τότε στο όνομα ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, διότι είναι έκτακτη ανάγκη, διότι πλήττεται η υγεία των ανθρώπων από τις εισόρευσεις χώρων, από αποβλήτων σε χώρο που δεν πρέπει, τότε πάμε σε λύσεις, ε, να μην πω την έκφραση, άντε να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το πρόβλημα της υγείας. Ενώ είναι μια, ε, μια χρονίζουσα κατάσταση δεν γίνεται με σωστό τρόπο και παραβιάζεται και κοινοτική οδονοδικία. Δεν σας κουράζω περισσότερο. Η τελευταία παρατήρηση και έχετε πιστεί πράγματι και για τη σοβαρότητα του θέματος είναι ότι περιοριστήκαμε λίγο ή περισσότερο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τη στενή έννοια. Η γνώμη μου είναι η εφαρμογή σωστής οδηγίας θα έχει και έχει οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη και για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τα ευρωπαϊκά κράτη και για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι μια διάσταση που πρέπει να την κουβεντιάσουμε. Έχει και τέτοιες διαστάσεις. Διότι οι παραβιάσεις πολλές φορές στοιχίζουν ε, και ερχόμαστε εκ των υστέρων να αναπληρώσουμε το κενό με πολλαπλάσιο κόστο κτλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Κουντή. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη. Α, παρακαλώ πάρα πολύ όμω, γιατί έχουμε μόνο 10 λεπτά για την επόμενη. Ε, θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα μπορούσαν να υποθούν διάφορα, αλλά προχωρούμε πηγόντω με την ελπίδα ότι θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό ε, κείμενο που μας ήρθε από την Κομισιόν ε, και που μας αφορά άμεσα ως Επιτροπή να προχωρήσουμε στην, στο νούμερο 22 που αφορά μια αναφορά της κυρίας Ντενίζα Λαστόφκοβα για την ενεργειακή βιομηχανία στην Σλοβακία. Και επειδή έχουμε μεταπράστια μέχρι τις 10 και, και μισή, παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Ε, η αναφέρουσα. Áno, ďakujem. Dobrý deň. Ε, na úvod by som chcela poďakovať všetkým e, za túto príležitosť. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που μου δίνετε τη δυνατότητα ε, να συμμετέχω προσωπικά σε αυτήν την συζήτηση της αναφοράς, την οποία έχουμε ήδη υποβάλει. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω την ε, αναφορά πρώτα. In a few words. Ε, ναι, μια ολιγόλογη παρουσίαση, αν μπορείτε. Λοιπόν, η αναφορά μας αφορά το σχέδιο παροπλισμού ε, του πυρηνικού εργοστασίου της ε, Γιασλόφς και Μπουχούνιτς ε, στην Σλοβακία. Θα ήθελα εγώ να εστιάσω την προσοχή μου σε τρία σημαντικά κατά την άποψή μας ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον προβλησμό τέτοιων πυρηνικών εργοστασίων. Ε, κοιτάξτε, η πυρηνική ασφάλεια ε, είναι πάρα πολύ ε, σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Δηλαδή ότι σε περιπτώσεις παροπλισμών η ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει και να συμμορφούνται με τα υψηλότερα δυνατά στάνταρ προστασίας. Και στην προκείμενη περίπτωση βεβαίως ο πλεισμός θα πρέπει ε, να ε, αναλυθεί ε, και να διεξαχθεί από εταιρείες οι οποίες να έχουν πιστοποιημένη γνώση του αντικειμένου. Ε, ασφάλεια λοιπόν ε, πρώτα και ε, γνώση των πυρηνικών θεμάτων. Αυτό ήταν το δεύτερο ζήτημα. Το τρίτο είναι η απαραίτητη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή έτσι ώστε ο παροπλισμός ε, να γίνει με σωστό τρόπο. Ε, οι παροπλισμοί τέτοιων πυρηνικών εργοστασίων δεν μπορεί να θεωρηθούν μικρά τοπικά προγράμματα. Και επομένως και η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι η προσήκουσα. Το εργοστάσιο στο οποίο αναφερόμαστε, στο Γιασλόφς και Μπουχούνιτσε, παροπλίζεται λόγω των απαιτήσεων της ένταξης της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την Σλοβακία έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτόν τον παροπλισμό. Ε, όμως εντωμεταξύ ε, συνέχισε η λειτουργία αυτού του πυρηνικού ε, εργοστασίου. ενώ ε, η Σλοβακία συνέλεγε χρηματοδοτήσεις ας πούμε για, την, ε, για τον ε, παροπλισμό. Μέχρι τώρα δεν έχουν μαζευτεί αρκετά χρήματα έτσι ώστε να ξεκινήσει ομαλά και να μπορέσει να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία παροπλισμού. Η Σλοβακία αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται στη φάση της αποξύλωσης. Ε, είναι αυτό που ονομάζουμε φάση φυσικού παροπλισμού. Και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το σχέδιο αυτό έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Το κονσόσιουμ, ε, το οποίο, η οργάνωση δηλαδή, την οποία εκπροσωπώ, αυτό το κονσόσιουμ για την ενέργεια, ζητά επισταμένως κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ βλέπουμε ελληματική συμπεριφορά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει καταβάλει μονάχα το 1 τρίτο του αναμενόμενου χρηματικού ποσού. Περιμένουμε λοιπόν ε, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ε, υπολείπονται από ένα συνολικό προϋπολογισμό 552, 553 σχεδόν εκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η συνέχιση ε, του ε, σχεδίου αυτού, η ασφαλής συνέχιση, ασφαλής και για το περιβάλλον και για τον ε, πληθυσμό. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η διαδικασία αυτή Εκτός από την ε, Σλοβενία, ε, Σλοβακία αυτή τη στιγμή ε, έχουν ξεκινήσει παροπλισμοί αντίστοιχοι και στην Λιθουανία και στην Βουλγαρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξακολουθήσουν τα προγράμματα αυτά να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να πω Ε, ότι από τη στιγμή που ο κύριος χρηματοδότης είναι ε, η Τράπεζα Ανασυγκρότησης ε, και το ΑΕΡΙΣ... πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης. Θα ήθελα να, μου, να σας προτείνω ενδεχομένως και αν μπορείτε να το δεχτείτε τη διοργάνωση μιας δημόσιας ακρόασης ή τέλος πάντων μιας διαβούλευσης για το θέμα αυτό. Για να συνοψίσω λοιπόν, ε, μιλάμε για τον παροπλισμό ενός πυρηνικού εργαστοσίου που έχει ήδη ξεκινήσει στη χώρα μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ε, η ικανοποιητική χρηματοδότηση έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σωστά η διαδικασία. Ευχαριστώ. Είναι η μετάφραση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κίρχνερ από μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Κίρχνερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου την αναφορά. Απαντώντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το πλαίσιο και το σκεπτικό της ε, επιπρόσθετης κρηματοδότησης ε, είναι βασισμένο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια και την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων. Είναι πλήρης ευθύνη των κρατών μελών και αυτό τι σημαίνει. <clears throat> σημαίνει και την ε, διασφάλιση επαρκών ε, κονδυλίων. Η Σλοβακία έχει δεσμευτεί να κλείσει το πυρηνικό εργοστάσιο αυτό στα πλαίσια της ανεμοθεσίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αντάλλαγμα δεσμεύτηκε να στηρίξει την Σλοβακική Δημοκρατία για τον παροπλισμό και όχι μόνο για τον παροπλισμό αλλά και για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες αυτού. Αυτή η δέσμευση ήταν μέχρι το τέλος του 2006. Τώρα υπήρξε ε, ξανά το τέλος, το τέλος του 2006 το ζήτημα του οικονομικού φόρτου όπως, και όπως προβλέπεται στο πρωτόκολλο της ε, προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίστηκε να δοθούν επιπλέον συμπληρωματικά κονδύλια, διότι το πρωτόκολλο δεν ήταν επαρκή σε νομική βάση πλέον. Συνεπώς, μέχρι το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 630 εκατομμύρια ευρώ προς τη Σλοβακία για τον παροπλισμό. Η αρχική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την ε, Σλοβακία δεν είχε πρόθεση φυσικά να καλύψει το πλήρες κόστος του παροπλισμού του εργοστασίου. Ωστόσο, εξαιτία της προόδου που έχει επιτευχθεί και επειδή ακριβώς η ασφάλεια είναι πρώτη στο ενδιαφέρον, αποφασίστηκε να επεκταθεί η χρηματική υποστήριξη πέρα από το 2013 και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ε, επιπρόσθετος 150 εκατομμύρια ευρώ ως οικονομική στήριξη από το 2014 έως το 2017. Αυτό μας κάνει συνολικά λίγο πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία καλύπτουν πάνω από το 50% του κόστους παροπλισμού. Έχει γίνει για το οποίο επίσης επανεκτίμηση του κόστους αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θεωρεί χρηματο, επαρκή χρηματοδότηση. Υπάρχουν τα κονδύλια και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι, δεν είναι μόνο το κόστος του παροπλισμού αλλά και το χρονικό πλαίσιο. Αυτά τα εργοστάσια πρέπει να κλείσουν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μας μένουν λοιπόν μόνο λίγα χρόνια μέχρι αυτό το χρονικό σημείο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικοί επίσης να μην δώσουμε παραπάνω χρηματοδότηση διότι έτσι θα βλάψουμε τον ανταγωνισμό. Τώρα, συμπερασματικά, για όλους αυτούς τους λόγους η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν έχει στόχο να καλύψει το πλήρες κόστος του παροπλισμού αυτό είναι στην ευθύνη της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η διασφάλιση δηλαδή των ε, κονδυλίων που λείπουν, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο παροπλισμός. Και τα κονδύλια αυτά, τα ευρωπαϊκά, ε, αποδοσμεύονται όταν χρειάζονται. Αυτό ήταν και μία εξάντε προϋπόθεση που είχαμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή η διάταξη, όπως και οι υπόλοιπε, εναρμονίζονται πλήρως με τις συστάσεις που έχουμε λάβει στα πλαίσια και του ελέγχου από το Ελληνικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κίρχνερ. Ο κύριος Πάσκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητοί ε, αναφέροντες, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι της Επιτροπής. Πρέπει να σας πω ότι το εργοστάσιο έκλεισε λίγο μετά τη γενική αναδιάρθρωση του όλου συστήματος από τη Westinghouse. Τότε ήμουν στη Σλαυκική κυβέρνηση όταν έγινε αυτή η αναδιάρθρωση και η ανοικοδόμηση και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, άρα πρέπει να ε, έχουμε υπόψη μας τα στοιχεία αυτά και υποτίθεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει 30 χρόνια ακόμη το πυρηνικό εργοστάσιο, αλλά επειδή μας το ζήτησε η Αυστρία, ε, συμφωνήσαμε να το κλείσουμε, δεν εμπιστεύονταν ε, οι αυστριακοί εταίροι την τεχνολογία του πυρηνικού εργοστασίου και μας ζήτησαν γι' αυτό το λόγο να μειώσουμε το χρόνο λειτουργία του πυρηνικού αυτού εργοστασίου. Παρά το ότι λειτουργούσε μια χαρά. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι θα παροπλήσουμε σταδιακά το πυρηνικό αυτό εργοστάσιο και φυσικά και δεν αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος. Είναι όμως ε, αμετάκλητη αυτή η διαδικασία, δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε, δεν μπορούμε να αναστείλουμε ε, τις εργασίες γιατί αυτό θα θέσει σε κίνδυνο και την ασφάλεια των πολιτών, όχι μόνο της Σλοβακίας αλλά και της Αυστρίας. Πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν ε, η αποξύλωση, ο παροπλισμός αυτού του πυρηνικού εργοστασίου. Βέβαια, εμεί είμαστε σε ένα διαφορετικό στάδιο σε σχέση με άλλου πυρηνικού σταθμού που παροπλίζονται. Το θέμα είναι όμω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε ε, τι εργασίε. Οι αρχικέ εκτιμήσει ε, τη Κομισιόν δεν είχαν υπολογιστεί με, έναν, ε, με το σωστό συντελεστή. Αν ε, συγκρίνεται τον ε, συντελεστή, παραδείγματο χάρη τη Λετωνία, δεν είναι το αντίστοιχο αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει. Βέβαια, εμεί θα συνεχίσουμε τα έργα για τον παροπλισμό, αλλά χρειάζεται τακτική χρηματοδότηση, στην οποία πρέπει να βασιζόμαστε, να μπορούμε να βασιστούμε. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην ε, Κομισιόν που λέει θα σας δώσουμε ένα ποσό συγκεκριμένο, μετά μας δεν θα μας το δώσει καθόλου. Και ο κύριος Φωνορομπάη ε, στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου είπε και αυτό στην απόψή του και πρότεινε να αυξηθεί στα 200 εκατομμύρια το ποσό από τα 100 εκατομμύρια. Άρα και το Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση από πλευράς Κομισιόν για το κόστος. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου. Ďakujem pekne. Veľmi, Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί ο συνάδελφος Πάσκα είπε τα πιο σημαντικά. Στηρίζω βέβαια την αναφορά αυτή και πιστεύω ότι αξίζει να τη στηρίξουμε για δύο λόγους πρέπει κανείς ε, να καταλάβει ότι όλα αυτά συμφωνήθηκαν ε, την στιγμή της ένταξης της Σλοβακίας. Ε, πριν την ένταξη λοιπόν η Αυστρία, η γειτονική μας χώρα, ζήτησε, απέτησε μάλλον αυτόν τον όρο που βεβαίως δεν ήταν εκείνη τη στιγμή απόλυτα επιτεύξιμος και βεβαίως έβαλε και τη Σλοβακία σε μία ε, θέση κατά κάποιο τρόπο αμυντική ε, και ε, γιατί εκείνη τη στιγμή η Σλοβακία ήθελε βεβαίως να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι ο χρόνος ζωής θα έπρεπε να ήταν τριακονταετής και όχι τόσο σύντομος. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός επίσης ότι με, όλα αυτά φτάσαμε σε έναν απαροπλισμό ο οποίος κρατάει περισσότερο, ο οποίος είναι πιο ε, ακριβώς, κοστίζει και περισσότερο γιατί ο τρόπος που επελέγει είναι ακριβότερος ε, και βεβαίως ε, και μέσα στα πλαίσια της ενεργειακής ε, πολιτικής ε, της Ατζέντα 2020 υπάρχουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις και όσο γίνεται πιο, όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί ο παροπλισμός, τόσο πιο χαμηλά είναι τα κόστη. Αυτό το ξέρουμε. Στην προκείμενη περίπτωση η Σλοβακία αναγκάζεται να ε, δαπανίσει περισσότερα χρήματα γιατί ο παροπλισμός διαρκεί ακόμα πέντε χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όσο πιο σύντομα ολοκληρωθεί ο παροπλισμός τόσο καλύτερα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Τσάλα. Η κυρία Άουκεν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αναφορά. Πριν από λίγο συζητήσαμε για την οδηγία ΕΠΕ και ακούσαμε και τα όσα μας απήντησαν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, βλέπουμε ότι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν βεβαίως και από ένα πυρηνικό εργοστάσιο αλλά ε, και ε, κίνδυνους, κίνδυνους μπορεί να παρουσιάσει και μια αγροτική εκμετάλλευση βεβαίως του των αναλογιών πάντοτε. Τώρα, αν μια χώρα επιλέξει να χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια, ε, είναι δικαίωμά της, ε, αλλά τα απόβλητα ε, και ο τρόπος με τον οποίο ξεφορτώνεται κανείς τα απόβλητα αυτά και ο τρόπος ο οποίος παροπλίζεται μια τέτοια εγκατάσταση είναι μια άλλη συζήτηση. Όταν η Κομισιόν είπε ότι θα μπορούσε ας πούμε να αντιπροσωπεύσει αυτή, ε, αυτό το εργοστάσιο ε, πρόβλημα στον ανταγωνισμό. Τι να σας πω, το πρόβλημα είναι ότι ωραία παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις αλλά δεν έχουμε ποτέ μία σαφή εικόνα του κόστους πρώτα ε, αναφερόμαστε και σκεφτόμαστε τις ενδεχόμενες τρευλώσεις του ανταγωνισμού και μετά λέμε πόσα χρήματα θα κοστίσει το να πάρουμε την α ή τη β απόφαση και να κάνουμε τη μία ή την άλλη λύση. Ε, και είναι γεγονός ότι υπάρχουν σε πολλές χώρες πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις ασφάλειας. Συμφωνώ λοιπόν με το θέμα αυτό της Σλοβακίας, αλλά θα πρέπει να αποσαφινιστεί ότι η Κομισιόν ήταν υπερβολικά ε, απλόχερη όσον αφορά ε, την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι ένα πυρηνικό εργοστάσιο ε, προκαλεί την ίδια μόλυνση με ένα χειροστάσιο. Θα πρέπει να τηρηθούν αυτές οι αναλογίες. Er Κοιτάξτε, ε, μήπως ε, κάποια χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν άμεσα για την ενέργεια αλλά για κάποιους άλλους λόγους. Εν πάση περιπτώσει Τώρα παραμένει το πρόβλημα του παραπλησμού ε, του εργοστασίου αυτού. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο παραπλησμός αυτός. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τις υποσχέσεις που δόθηκαν στην ε, Σλοβακία. Από την άλλη πλευρά είναι σκανδαλώδες ε, το ότι ξεκίνησαν και δημιουργήθηκαν αυτά τα εργοστάσια χωρίς προβλέψεις και επίσης χωρίς καμία πρόβλεψη όσον αφορά το κόστος παροπλισμού τους και αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να το μάθουμε. Μία και καλή. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μαθητές σε αυτή την περίπτωση. Γιατί δεν πρέπει να επαναληφθούν αυτά τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, το κόστος παροπλισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται. Ο κύριος Γιάρ ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο του κύριου Γιάρ. Μάλιστα, θα προτείνω κι εγώ κάτι. Προτείνω λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά για τους εξής λόγους. Πρώτον, θέλουμε γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την ε, κοιτάξουμε. Έπειτα, χρειάζομαι Χρειάζεται να δούμε τους κανόνες, να έχουμε μια γενική εικόνα, να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσει, να δούμε τι γίνεται με τον ανταγωνισμό στις ε, περιπτώσεις ε, παροπλισμού ε, πυρηνικών εργοστασίων. Εντάξει, έχω τη γενική εικόνα, αλλά δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν είμαι εμπειρογνώμονας και έπειτα χρειάζεται να ορίσουμε επακριβώ το πρόβλημα, να δούμε τι γίνεται με τον υπολογισμό του κόστου στην Σλοβακία, τι μας περιμένει στο μέλλον και να δούμε τι έχει να πει η Επιτροπή για το πώς ε, θα ε, εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν η πρότασή μου είναι να περιμένουμε μέχρι το τέλος και μετά να ψηφίσουμε. Να αναφερθούν στο πρωτόκολλο αυτά τα πράγματα, γραπτή απάντηση, κανόνες ε, διαδικαστίας και σε κόστους από την Σλοβακία. Και μετά αυτό να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας έρθει απάντηση. Επομένως την κρατούμε ανοιχτή εκτιμώ βεβαίω ότι τέτοιου του ζητήματα υπερβαίνουν τα όρια τη επιτροπή Αναφορών. Uh, I not... Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να προωθήσουμε την αναφορά αυτή σε άλλες επιτροπές. Ενδεχομένως ακόμα και στον Ombudsman, τον διαμεσολαβητή, γιατί είναι διαφορετικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε να λύσουμε εμείς φυσικά. Χρειαζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες και από την Σλοβακική πλευρά και από την ε, ε, Κομισιόν ε, πρώτα. Αλλά φοβούμε ότι ως Επιτροπή Αναφορών δεν μπορούμε μόνοι μας να χειριστούμε το ζήτημα αυτό. Θα ακολουθήσω λοιπόν την πρόταση του κυρίου Γιάρα. Αναρωτιέμαι όμως ε, μάλλον όχι. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε επιπλέον στοιχεία και ενδεχομένως θα πρέπει να προωθήσουμε την αναφορά αυτή αλλού. Φρονώ ότι έχει υπάρξει εδώ ελλειπής τακτική όσον αφορά την ε, ασφάλεια αυτής της πυρηνικής εγκατάστασης. Και αυτοί, αυτές οι ελλείψεις αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Είδαμε τι έγινε μετά το Τσερνόμπιλ. Και τώρα φαίνεται ότι τα προβλήματα αυτά έχουν μετατοπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, και ενδεχομένως δεν θα πρέπει καν να είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων ζητήματα τέτοιου είδους, αλλά να περάσει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό το ζήτημα, ας πούμε, δεν απασχολεί, δεν, δεν αφορά μονάχα τη Σλοβακία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια γενική θεώρηση. Ε, θέτω κάποια γενικά ερωτήματα, δεν είναι απαραίτητο να απαντηθούν άμεσα. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να σκεφτούμε σε ποιες άλλες ε, επιτροπές μπορούμε να προωθήσουμε αυτήν την αναφορά έτσι ώστε να έχουμε και μια επιπλέον γνωμοδότηση. Αναρωτιέμαι. Now we go. Uh, you have to be thinking the issue. Το σκέφτεστε κύριε Μποστινάρου. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι Έκλεισε το μικρόφωνο, δυστυχώς. I did it, but uh, then he died. Πέθανε το μικρόφωνο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή πρέπει να είναι η Ήτρε, κατ' με, η οποία αντιμετωπίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια. Όμως, είναι σημαντικό να δούμε και ποιες είναι οι νομικές δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν τα έκανε η Σλοβακική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή που αποφάσισε να ζητήσει από τη Σλοβακία να κλείσει τον πυρηνικό αυτό σταθμό. Ακόμη και αν τότε η αξιολόγηση, η εκτίμηση ήταν ε, μη ρεαλιστική, αν είναι διαφορετικά τα νούμερα, θα πρέπει κάποιος να δει τις διαφορές μεταξύ της τότε εκτίμησης και της σημερινής πραγματικότητας και αυτό είναι σοβαρό. Βρισκόμαστε σε καιρό κρίση. Δεν μπορούμε απλά να ζητάμε από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, είτε αυτή είναι η Σλοβακία είτε άλλη χώρα, να λέω ότι είναι δική σας η ευθύνη να κάνετε αυτό και το άλλο. Και ποιος θα πληρώνει αυτά, η Σλοβακία, στην προκειμένη περίπτωση. Είμαι πολύ αντίθετος προς αυτή τη φιλοσοφία. Ήταν μια κοινή λύση την οποία προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Σλοβακία και θα πρέπει με ρεαλιστικό τρόπο να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Και βέβαια να γίνει και με λογικό τρόπο και να λήξει στο μότερο δυνατόν. Άρα καλό είναι να κάνουμε μια ρεαλιστική εκτίμηση των εξελίξεων και επαναλαμβάνω να ακούσουμε και την άποψη της Επιτροπής Ήτρε. Βέβαια, σίγουρα η Επιτροπή μας πρέπει να διατηρήσει ανοιχτή την αναφορά και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και ένα είδος προηγούμενου, γιατί φαντάζομαι ότι σύντομα θα έχουμε και τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες και στη Βουλγαρία και όχι μόνο. Και θα κληθούμε ως Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε και, άλλα, και αλλού αντίστοιχα προβλήματα. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, η πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Ε, we keep it open. We send... Ωραία, παραμένει ανοιχτή η αναφορά, την στέλνουμε στην Ήτρα και περιμένουμε και τα επιπλέον στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ. Περνάμε τώρα στην κανονική σειρά της ημερησίας διάταξης. ενώ στο σημείο 15 αναφορά της Τανιέλα Σπέρα Ιταλικής Ιθαγένειας. σχετικά με την κατασκευή ενός αγωγού αερίου στην Απουλία. Είναι εδώ η κυρία Σπέρα, αν δεν απατώμε. Sí. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ την Επιτροπή Αναφορών που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εδώ έτσι ώστε να παρουσιάσω αυτά τα προγράμματα ε, εξ ονόματος των πολιτών του Τάραντο μέσω της ε, Ένωσης ε, των ε, Ιωνίων Δεσμών, Ασοσιαστιών Ελεγκάμι Ιόνιτσι, είχα υποβάλει μια αναφορά η οποία αφορά το, το πρόγραμμα Τεμπαρόσα, ενώ η δεύτερη αναφορά μου αφορά ένα άλλο σχέδιο, ένα άλλο σχέδιο λοιπόν το οποίο είναι πιο εξειδικευμένο και αφορά ε, την ε, ε, ενδεχόμενη παραβίαση της ΕΠΕ από την εταιρεία ΕΝΗ. Στην, για την προκείμενη περίπτωση έχουμε υποβάλει και καταγγελία η οποία αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο βαραίνει πολύ την πόλη μας, την πόλη του Τάραντο και που ακόμα δεν έχει λυθεί με κανένα τρόπο θα ήθελα να διαβάσω μια ανακοίνωση σχετικά με το Παρόσα. γιατί εντωμεταξύ έχουν υπάρξει εξελίξεις. Έχουμε ε, βρει κάποια νέα έγγραφα και έχουμε πάρει κάποιες νέες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στην ίδια εισαχθήσα αναφορά. Λοιπόν, ε, είχαμε ε, αναφέρει παραβίαση ενδεχόμενη της οδηγίας ε, ΣΕΒΕΖΟ και της ε, οδηγίας ΕΠΕ. Όσον αφορά τώρα τις ε, τις ε, εν λόγω οδηγίες ε, και όσον αφορά τις ενδεχόμενες παραβιάσεις πρέπει να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο οδηγίες προβλέπεται πρώτερη διαβούλευση όσον αφορά είτε δημιουργία είτε τροποποίηση υπαρχουσών εγκαταστάσεων κυρίως όσον αφορά την μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία. Ακόμα και από την περίοδο του σχεδιασμού θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιπτώσεων, καθώς επίσης και το ενδεχόμενο ε, ε, εναλλακτικών ε, λύσεων. Η διαδικασία ΕΠΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την αρχή της ασφαλείας. Οι πολίτες επίσης θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να, κάνουν, να γνωρίζουν πρώτον τους κινδύνους και να γνωρίζουν πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν σε περίπτωση κινδύνου. Το 2011 υπήρξε ένα κοινό διάταγμα από δύο Υπουργείο ε, και ε, μετά από παραγραφή των αποφάσεων για το 2009 και το 2008, ε, κυρίως όσον αφορά την περίπτωση πυρκαγιάς, ε, διαπιστώνουμε ότι ε, δεν έχουν ληφθεί υπόψη αυτού του είδους οι προβλέψεις βάσει της οδηγίας σε βέζο. Παρόλο που δεν εκαλύπτονται αυτές οι προδιαγραφές από την εν λόγω εγκατάσταση, οι Ιταλικές αρχές έδωσαν έδωσαν την σύμφωνη γνώμη τους. Σημειώνω ότι ε, εμείς σαν Ένωση ε, Λιγκάμι Ιόνιτσι είχαμε ήδη σημειώσει και είχαμε υποβάλει στην αρμόδια αρχή αναφορά ε, στην οποία ακριβώς αναφέραμε την μη συμμόρφωση της εταιρείας όσον αφορά αυτές τις ε, ε, αυτά τα σημεία. Επίσης, ε, εμείς δηλώσαμε ότι το κοινό δεν εγνώριζε την μη συμμόρφωση της εταιρείας. Σημειώσαμε επίσης ότι οι πληροφορίες προς το κοινό ήταν σαφώς ατελείς. Επομένως, δεν είχε το κοινό απαραίτητες πληροφορίες. Αυτές τις πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται από την οδηγία σε Βέζο. Βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας σε Βέζο, το κράτος μέλος δεν μπορεί να δώσει άδεια λειτουργίας εάν τα μέσα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη κινδύνου είναι ελλειπή. Επίσης και σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΠΕ είναι ελλειπής. Ε, υπενθυμίζω εδώ ότι εδώ μιλάμε για εγκατάσταση η οποία θα δημιουργηθεί στα πλαίσια υπάρχοντος διηληστηρίου. Επομένως, μιλάμε για μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη, η οποία σαφώς εμπίπτει στην οδηγία σε Βέζο. Επίσης, ε, ε, εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα, το οποίο, για ένα σχέδιο, συγγνώμη, το οποίο και έχει μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μπορεί να έχει επιπτώσεις στο, ε, στην υγεία. Το άρθρο 9 της Οδηγίας Εβέζο σαφώς και ρητά αναφέρει ότι θα πρέπει αμελητή, το τονίζω, αμελητή να στέλνονται όλα αυτά τα στοιχεία για την, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και για τις επιπτώσεις επί της υγείας. Αυτό δεν έγινε. Επίσης, όσον αφορά την συμμετοχή του κοινού, όσον αφορά την διαβούλευση, ούτε αυτή η προϋπόθεση έχει καλυφθεί. Επίσης και επιπλέον το κοινό δεν γνώριζε ότι υπήρχε μη συμμόρφωση της εταιρείας και ε, επομένως το κοινό δεν ήταν σε θέση, οι πολίτες δεν ήταν σε θέση να υποβάλουν οποιασδήποτε παρατηρήσεις νομίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ε, μία οποιαδήποτε ε, απόφαση η οποία δεν θα περιλαμβάνει ΕΠΕ και δεν θα περιλαμβάνει διαβούλευση ε, με τους πολίτες. Πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε εδώ για 180.000 κυβικά υγρού τα οποία θα διακινηθούν, ναι, ε, ε, ε, πέρα από αυτό λέω υπάρχουν και πάρα πολλοί κίνδυνοι όσον αφορά την υγεία του κοινού. Επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο αγωγός περνάει από έναν πολύ πυκνά χρησιμοποιούμενο δρόμο. Υπάρχει ε, κοντά και ένα ψυχαγωγικό πάρκο, ε, υπάρχει και ένα κέντρο παλαιό, ε, παλαιό νοσοκομείο, το οποίο είναι κέντρο υποδοχής ατόμων υπό αποτοξίνωση κτλ. Μιλάμε επομένω για μια περιοχή η οποία σε περίπτωση κινδύνου μπορεί να έχει αυτός ο κίνδυνος πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και επομένως ε, ε, εν προκειμένου πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ε, μια ΕΠΕ. Επίσης, εμείς έχουμε δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και γνωρίζετε επομένως όλα τα στοιχεία. Ευχαριστώ. παρακαλώ από τη μεριά της Κομισιόν η κυρία Μίκυλσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανοίξει EU Pilot για τις δύο αυτές αναφορές και έχει στείλει και διάφορε επιστολέ στι Ιταλικές Αρχέ στη διάρκεια του του, συγγνώμη, του προηγούμενου έτους συγκεκριμένα. Τρει επιστολέ, τρει απαντήσει λάβαμε. Η τελευταία είναι τη 14η-15η Ιανουαρίου, άρα τη μελετούμε ακόμα. Μπορούμε να σα δώσουμε όμω κάποια στοιχεία σε σχέση με τις εικαζόμενες παραβιάσεις της ε, νομοθεσίας. Επαναλαμβάνω, κάποιες τις εξετάζουμε ακόμη. Σε ό,τι αφορά την ε, αναβάθμιση, στον εξονισμό του δηληστηρίου, στις 27 Οκτωβρίου του 2011 δόθηκε η έγκριση μέσω ενός διατάγματος ε, στο οποίο ορίζονται το πώς θα λάβουν χώρα δημόσιες διαβουλεύσεις. Τελευταία γίνεται τον Ιανουάριο του 2011 Επίσης υπήρχε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ε, μία μη τεχνική σύνοψη της ε, ΕΠΕ. Στην οδηγία ΕΠΕ λέγεται ότι αναλυτικές διευθετήσεις για την ενημέρωση του κοινού και τη διαβούλευση με αυτό καθορίζονται από τα κράτη-μέλη. Επίσης αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης λαμβάνονται υπόψη για την ε, ανάπτυξη και την εξέλιξη της δικασίας ε, έγκρισης, ε, consent. Στην περίπτωση αυτή δεν δόθηκαν νομοδοτήσεις μετά από τις δύο διαβουλεύσεις με το κοινό. Και αναφέρεται στην οδηγία επέτη, περιεχόμενο θα πρέπει να καλυφθεί, αλλά εδώ γίνανε επιδημιολογικές μελέτες και μελέτες ανάλυσης κινδύνου που δεν συμπεριλήφθησαν όμως δεν μπορούμε να ορίσουμε παράβαση οδηγίας ΕΠΕ τώρα. Σας έχουμε στείλει μια γραπτή ανακοίνωση και εξακολουθεί να είναι το project στη φάση του σχεδιασμού, άρα δεν μπορούμε τώρα να παρατηρήσουμε κάποια παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ. Επίσης, στην αναφορά εντοπίζεται η καζόμη παραβίαση της οδηγίας για την ασφάλεια των τροφίμων. Θέλετε να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί ε, στην παρουσίαση σας σήμερα δεν ε, το θίξετε αυτό το θέμα. Θέλετε? Άρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, την Καματαλήτα Σάνκο. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες και μετά εγώ θα περάσω στις καζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας σε Βέζο. Ευχαριστώ πολύ. Πάλο Καρικάτο από την DG Sanko. Στην ε, αναφορά την οποία έχουμε λάβει και στα ε, ε, συνοδεύοντα έγγραφα πληροφορούμεθα ότι στην περιοχή δίπλα στο δηληστήριο υπάρχουν καλλιέργειες ε, ε, διθύρων ε, μαλακίων. Αυτού του είδους οι καλλιέργειες και αυτά τα προϊόντα σαφώς υφίστανται τις δεσμεύσεις της λεγόμενης δέσμης υγιεινής που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2007 το άρθρο 2, τμήμα 7 του παραρτήματος 3, ορίζει ποιες είναι οι απαιτήσει και προϋποθέσεις παραγωγής και συλλογής των των ε, μαλακίων και επίσης καθορίζει τα χαρακτηριστικά των ζωνών παραγωγής. Επίσης, στο άρθρο 2 του παρατήρηματος 2 του 854 ε, συγγνώμη, ε, ορίζει τους επισήμους ελέγχους που θα πρέπει να κάνουν οι τοπικές αρμόδιες αρχές ε, στις ζώνες παραγωγής. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση καθώς επίσης και τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται από τις αρμόδιες αρχές στις ζώνες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των επιδημιολογικών αναλύσεων ε, που θα πρέπει να διενεργηθούν από τις αρμόδιες αρχές αρμόδιες αρχές υγιεινής, προστασίας της υγείας κτλ. Ε, προτού αποφασίσουν να κατηγοριοποιήσουν μια περιοχή ως εγκεκριμένη ζώνη παραγωγής ζώντων μαλακίων. Αυτό σημαίνει ότι μια ζώνη παραγωγής ζώντων μαλακίων είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Είναι ε, μία διαδικασία η οποία θα πρέπει με προσοχή να αντιμετωπιστεί και μάλιστα και με μεγάλη αίσθηση ευθύνης από τις εθνικές τοπικές αρχές υγιεινής. Οι αρμόδιες λοιπόν αρχές υγιεινής όταν αποφασίζουν να κατηγοριοποιήσουν ε, μια περιοχή ως συγκεκριμένη ζώνη παραγωγής μαλακίων θα πρέπει να λάβουν υπόψη και να συνυπολογίσουν όλους τους παράγοντες μόλυνσης. Δεν πρέπει δηλαδή να περιοριστούν σε έναν μικροβιολογικό έλεγχο των υδάτων, ας πούμε, αλλά θα πρέπει να λάβουν υπόψη και την ενδεχόμενη παρουσία χημικών, τοξικών ε, ουσιών κλπ. πριν αποφασίσουν ότι η ζώνη αυτή μπορεί να θεωρηθεί η εγκεκριμένη ζώνη παραγωγής μαλακίων. Έχω έχω λάβει ε, τα έγγραφα από την συνάδελφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Μελετώντας τα λοιπόν, διεπίστωσα ότι η ζώνη ε, παραγωγής έχει κλείσει λόγω ε, παρουσίας επικίνδυνων τοξινών, διοξίνης κτλ. ήδη από το 2011 μετά από απόφαση του Δημάρχου του Τάραντο. Εάν κατάλαβα καλά λοιπόν, αυτή η περιοχή τούτη τη στιγμή δεν ε, ε, παράγει πλέον ζώντα μαλάκια, διότι ο Δήμαρχος ε, αποφάσισε ότι υπάρχει εμφανής μόλυνση της, των καλλιεργούμενων μηδιών. Όμως, μία τέτοια περιοχή δύσκολο θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί ως εγκεκριμένη ζώνη παραγωγής ε, των μαλακίων, ούτως ή άλλως. Αυτό που θέλουμε να αξιολογήσουμε και για την ώρα δεν έχουμε ακόμα λάβει αρκετά στοιχεία ή έγγραφα, αυτό που πρέπει λοιπόν να ε, διακριβώσουμε είναι ποιες ήταν οι παράμετροι και οι ε, διαδικασίες ε, ε, κατηγοριοποίησης της Μάρε Πίκολο πριν από το 2011. Γιατί τώρα ξέρουμε ότι μετά την απόφαση του 2011 η ζώνη έχει κλείσει, δεν παράγει πλέον ζώντα μαλάκια και επομένως δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα διατροφικό, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί φαντάζομαι ότι φυλάσσεται κιόλας η περιοχή, δηλαδή υπάρχει μια φύλαξη έτσι ώστε να μην συνεχίζεται η παραγωγή μαλακίων αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησαν οι τοπικές αρχές της Απουλίας έτσι ώστε να κατηγοριοποιήσουν αυτή την περιοχή ως συγκεκριμένη ζώνη παραγωγής πριν το 2011. Σε αυτή την κλειστή περιοχή ε, υπάρχουν ε, αυτά τα μικρά ε, μύδια τα οποία ε, ακόμα δεν μπορούν να, να καταναλωθούν, δεν είναι βρόσιμα ακόμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, πώς να σας το πω λέει ο μιλητής, είναι σαν τα μικρά μυδάκια. Επομένως, υπάρχουν εκεί υπάρχουν εκεί γόνια, στο πούμε, μηδιών που θα πρέπει να ελεγχθούν και για τη διοξίνη και για άλλα ε, τοξικά ε, ε, στοιχεία. Ε, ενδεχομένως λοιπόν, εάν είναι δυνατόν, αυτά τα νεογνά θα πρέπει να μεταφερθούν σε μια άλλη καθαρή περιοχή, έτσι ώστε εκεί να μεγαλώσουν. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω λοιπόν τώρα μιλώντας για τι εικαζόμενε παρεμβάσει Οδηγίας ΕΒΕΣ. Όπω σα είπα, στείλαμε τρει επιστολές στις ταλικές αρχές πήραμε και τις απαντήσεις τους αυτό που μπορούμε ήδη να συναγάγουμε και μπορώ να σας δώσω τις σχετικές πληροφορίες που μας έδωσαν τελικές αρχές είναι, όπως μας είπαν λοιπόν, η εκτίμηση της προκαταρκτικής έκθεσης ασφάλειας ε, και της σχετικής μελέτης, ε, προκαταρκτικής μελέτης ε, σκόπιμότητας υπευλήθη στις 27 Μαρτίου του 2012, όμως υπήρξε αναστολή της ανάλυσης για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δημόσιες διαβουλεύσεις, να αναλυθούν τα συμπεράσματα και μετά να μπορέσουν οι αρχές να, αποφασίσουν για τις δραστηριότητες με βάση τις εξελίξεις. Στις 30 ε, Αυγούστου λοιπόν ο Δήμος του Τάραντο ζητεί από το Φορέα Εκμετάλλευσης να δημοσιεύσει νέες ε, ε, ανακοινώσεις και ενημέρωση του κοινού. Υπήρχε λοιπόν αναστολή, όπως είπα, της αξιολόγησης της έκθεσης ασφάλειας. Οι αρμόδιες αρχές δεν είναι λοιπόν μέχρι τώρα σε θέση να συντάξουν ένα νέο εξωτερικό ε, σχέδιο ε, της ανάγκης, ούτε να εκπληρώσουν τις απαιτήσει για την ε, αναγνώριση κάποιων παρενεργειών ντόμινων, θέλετε όπως προβλέπετε στην οδηγία σε Βέζο. Υπάρχει όμως ένα προσωρινό, ένα προκαταρκτικό σχέδιο το οποίο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011 και το οποίο συμμορφούνται προς τις γενικές κατευθύνσεις ε, για τα emergency αυτά plans. Οι αρχές επίσης μας είπαν ότι ένα νέο σχέδιο ε, έκτακτης ανάγκης θα καταρτιστεί, θα γίνουν και οι δημόσιες διαβουλεύσεις και θα αξιολογηθούν οι τυχόν ε, επιπτώσεις, ε, παρεμπιπτώσεις επιπτώσεις. Και μετά θα δοθεί η άδεια σκοπιμότητας. Καταλήγουμε λοιπόν ε, στα εξή συμπεράσματα. Ναι, με αναληθεύει ότι οι πληροφορίε τη έκθεση ασφάλεια είναι πολύ σημαντικέ για την κατάρτιση εξωτερικών σχεδίων έκτακτη ανάγκη ε, και τον καθορισμό των διαφόρων επιπτώσεων. Φαίνεται όμως ότι οι αρχές έχουν μάλλον στα χέρια τους ήδη τις πληροφορίες που χρειάζονται η μόνη πληροφορία που τους λείπει είναι τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων. Τίθεται επίσης το θέμα κατά πόσον ε, το κοινό έχει ε, δώσει τη γνώμη του ή έχει υπάρξει επαρκής διαβούλευση με το κοινό. Στείλαμε μια επιστολή ε, το Δεκέμβριο του 2012 <coughs> Μα απάντησαν ε, οι Ιταλικέ αρχέ στι 14 και 15 Ιανουαρίου. Μελετούμε την απάντησή τους, οπότε σύντομα θα συντάξουμε μια γραπτή ανακοίνωση που θα στείλουμε στην Επιτροπή Αναφορών και θα σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα ε, των ερευνών μας και στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη αναφορά... Μπορείτε να είστε λίγο πιο σύντομοι, επειδή έχουμε κι άλλε πολλέ αναφορέ αν είναι δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δύο αναφορές ε, τις εντάξαμε στον ίδιο φάκελο. Δεν έχουμε εντοπίσει παράβαση της ε, νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για την πρώτη αναφορά. Για τη δεύτερη αναφορά όμως που ήσασταν πιο συγκεκριμένοι και εκεί ε, μας αναφέρετε για τέσσερα διαφορετικά project καζόμενες παραβιάσεις, πρέπει να σας πω ότι οι αρχές τους ζητήσαμε τουλάχιστον να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Λάβαμε κάποιες, ε, αλλά με αυτές δεν στοιχειοθετείται παράβαση. Κανένα από τα τέσσερα project μας αναφέρατε. Για να είμαστε σύντομοι, ε, μπορώ να σας πω ότι θα σας δώσουμε εγγράφος ε, τις απαντήσεις πολύ σύντομα, αν συμφωνείτε, τα σχετικά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει την επικοινωνία της με την Κομισιόν. Η κυρία Άουκεν ζήτησε το λόγο. Just briefly, uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Φυσικά να το κρατήσουμε ανοιχτό. Σοκαρίστηκα όταν άκουσα αυτά που είπατε, πως ε, αυτά τα μύδια προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Δηλαδή, έλατε τώρα, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να, να, να καταλήγουν στο, στο νερό. Δεν είναι απαραίτητο να ε, απαγορεύεται να, να, να καταλήγουν στα μύδια. Αυτά πέφτουν στη θάλασσα, πέφτουν στο περιβάλλον και συγκεντρώνονται τοξικές ποσότητες και πρέπει να ανησυχείτε για το ότι η συγκέντρωση είναι ε, ίδια στα μικρά μύδια όσο και στα μεγάλα. Ευχαριστώ κύριε ε, Αουκένο. Κύριος Γιάρ παρακαλώ. Μίστερ Γιάρ. Thank you. Και εγώ συμφωνώ, θα ήθελα να αφήσουμε την ε, αναφορά ανοιχτή μέχρι να πάρουμε την γραπτή ανακοίνωση της Επιτροπής. Αφού μας λένε και όλες ότι βρίσκονται στη διαδικασία σύστασή της. Να δούμε μετά τι γίνεται με τα μύδια. Φυσικά και είναι επικίνδυνη η διοξίνη. Δεν ε, είναι μόνο τα μύδια, υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν εκεί πέρα. Δεν απαραίτητο τα φάμε δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ συμφωνώ να μείνει η αναφορά ανοιχτή. Ε, κρατούμε την αναφορά ανοιχτή και προχωρούμε στην επόμενη. Ε, παρακαλώ τον κύριο Σέργιο Ντιάννα να την παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και το έγκριτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δέχτηκε την αναφορά μας. Ah, Υπάρχει και ο αριθμός 16. Ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος. Μα έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και του 16. Δεν είναι δικό μου το λάθος, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, παρακαλώ κύριε Διάννα, έχετε το λόγο. Ehm, ma c'è la 17, e la nostra è la 18. Η δικιά μα είναι η 18 όμω. Υπάρχει ακόμα η 17. Ci siete prima voi. Ε, allora, ε... Εντάξει λοιπόν, καλή σας μέρα. Εγώ είμαι εδώ για τρεις αναφορές. Την 483 του 2007, για την 1147 ε, του 2008, καθώς επίσης και τη 1472 του 2009. Ε, ως εκπρόσωπος όλων των υπαλλήλων. Λοιπόν, οι τρεις αναφορές αυτές αφορούν ένα προβλεπόμενο τερματικό σταθμό ε, ε, επανεριοποίησης ε, στον κόλπο της εταιρείας της και αναφέρομαι κυρίως σε θέματα ασφαλείας τα οποία τίθενται ένα αμφιβόλο βάσει αυτών των σχεδίων. Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, πρέπει να σας πω ότι πρώτα απ' όλα πρόκειται για, ένα, ε, για μια μονάδα επανεωροποίησης ε, στο λιμάνι της Τεριέστης από την Ισπανικών Συμφερόντων Gas Natural, ε, καθώς επίσης και μια offshore στον κόρπο της Τεριέστης από την Αίωνα. Όσον αφορά τα δύο πρώτα σχέδια μετά από την πρόσφατη παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ιταλίας έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ΕΠΕ λόγω ελήψεων που το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ε, ε, ε, διακριβώσει. Παρότι το ίδιο το Υπουργείο είχε δώσει το πράσινο φως αρχικά θα πρέπει να υπάρξει και μια ΕΠΕ όσον αφορά το ε, άλλο σχέδιο το οποίο ε, αφορά δηλαδή την προβλήτα στην ε, την εγκατάσταση στη θάλασσα, στον κόλπο της ταιριές της. Πρέπει να πω ότι ότι η μονάδα στον κόλπο της Τεριέστης έχει λάβει αδειοδότηση μετά από χωριστή διαδικασία ΕΠΕ. Δηλαδή ε, πρώτα ε, ε, αδειοδοτήθηκε η μονάδα επανεριοποίησης και μετά με ξεχωριστή διαδικασία ο αγωγός σύνδεσης. Και εδώ βεβαίως έχουμε κατάφορη παραβίαση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο αυτής της μονάδας επανεριοποίησης στην Τεριέστη έχει ε, αδειοδοτηθεί, πρέπει να σας πω, χωρίς ε, την στρατηγική ε, αξιολόγηση η οποία είναι απαραίτητη όταν, όπως συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση, γίνονται τροποποιήσεις στο συνολικό ρυθμιστικό σχέδιο του λιμανιού της Τεριέστης. Στην προκείμενη περίπτωση όμως ακόμα τώρα δεν έχουμε στρατηγική αξιολόγηση. Αυτά τα ε, σχέδια για μονάδες ε, επανεριοποίησης ε, πρέπει να σας πω ότι αφορούν τρεις χώρες, την Ιταλία, την Κροατία και τη Σλοβενία και όχι μονάχα μία. Δύο εκ των οποίων είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το, το τρίτο βρίσκεται πρώτων θυρών. Ε, όλοι, όλα τα σχέδια αυτά αφορούν τον κόλπο της εταιριές της και οπωσδήποτε θα πρέπει να υποστούν την διασυνοριακή στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέχρι τώρα εμείς έχουμε διαπιστώσει παραβιάσεις της ε, κοινοτικής νομοθεσίας ήδη σε αυτή τη φάση και επομένως φρονούμε πως δεν πρέπει να περάσουν τα σχέδια αυτά στην επόμενη φάση όλα τα απαραίτητα ε, έγγραφα θα πρέπει να κοινοποιηθούν ε, και στην Σλοβενία. Η κατάσταση λοιπόν είναι όπως σας την περιγράφω. Όσον αφορά το θέμα της ασφαλείας και τα δύο ε, σχέδια βεβαίως οδηγούν σε αύξηση ε, των ε, κινδύνων της ναυσιπλοείας στον κόλπο της της. Ε, όσον αφορά δε το σχέδιο της ε, Gas Natural, ε, πρέπει να πω ότι εγκαθίσταται στο βιομηχανικό πάρκο της Τεριέστης με αποτέλεσμα να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο για τον αστικό ιστό της πόλης της Τεριέστης. Επομένως, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση και όσον αφορά την οδηγία σε Βέζο για βιομηχανικούς κινδύνους, κυρίως όσον αφορά την εγκατάσταση στο λιμένα, το on-shore, όχι το off και βεβαίω να προβλεφθεί διαβούλευση με, ε, με τον ενδιαφερόμενο πληθυσμό. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δεν έχει λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση ο κόσμο έτσι ώστε να αξιολογήσει ε, το, ε, ε, τα σχέδια αυτά, κυρίως τα σχέδια της ε, εταιρείας Gas Natural στο λιμάνι της Τεριές της. λοιπόν πληροφόρησης, η οποία διαπιστώνεται σε ολόκληρη τη διαδικασία ΕΠΕ. Τα σχέδια αυτά, τα οποία πρέπει να πω ότι είναι παράλογο να υποβάλλονται για τον κόλπο της ταιριές της έχουν απόσταση 15 χιλιόμετρων περίπου το ένα από το άλλο ε, και αναφερόμαστε ε, σε εγκαταστάσεις οι οποίες, από τις οποίες θα περνούν 8 δισεκατομμύρια κυβικά ε, αερίου κάθε χρόνο και επομένως κατανοείται ότι πρόκειται για νούμερα τρομερά και παρόλα αυτά βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης αυτά τα σχέδια θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση ε, και των ε, κινδύνων τρομοκρατικών χτυπημάτων που μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα και για τον τοπικό πληθυσμό αλλά και για την αυσιπλοεία. Όσον αφορά τον κόλπο της ε, Τεριέστης, εδώ και 40-50 χρόνια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε έναν από τους ε, πιο σημαντικούς ε, τερματικούς ε, πετρελαϊκούς σταθμούς της Ευρώπης. Εάν δημιουργηθεί και ο τερματικός σταθμός του αερίου της Gas Natural, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος λόγω κυτνίασης με την υπάρχουσα πετρελαϊκή εγκατάσταση. Και βεβαίω σε περίπτωση προβλήματο ε, υπάρχει το ενδεχόμενο να μπλοκαριστούν ε, οι μεταφορές πετρελαίου προς την Ευρώπη. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι και τα δύο σχέδια θα οδηγήσουν σε αύξηση της ατμοσφαιρικής ε, ρήπανσης σε μία περιοχή όπως είναι το Φρίουλι Βενέτσια Τζούλια, που ήδη, ε, για την οποία ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιπαραβάση ήδη από το 2008 ακριβώς όσον αφορά το θέμα της ποιότητας ε, του αέρα που βεβαίως θα επιβαρυνθεί περαιτέρω ε, μετά από την ε, δημιουργία αυτών των εγκαταστάσεων. Και φυσικά στην ΕΠΕ δεν έχει ουδόλως ληφθεί υπόψη το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο σημείο το οποίο κατά την άποψή μας είναι σημαντικό. Η διαδικασία ΕΠΕ προβλέπει την πρόταση εναλλακτικών σημείων στην περίπτωση της εγκατάστασης επαναεριοποίησης ε, δεν έχει ε, καθόλου ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή. Ε, από την αρχή είπαν ότι θα γίνει μία εγκατάσταση στο λιμάνι της Τεργέστης και άλλο ένα offshore 400 μέτρα από την Αιγελίτιδα ζώνη της Σλοβακίας. Τελευταία σκέψη η οποία είναι πολύ σοβαρή κατά την άποψή μας, μια και μιλάμε ε, για διασυνοριακού ενδιαφέροντος ε, θέμα ε, και που επομένως θα πρέπει να εφαρμοστούν εδώ οι διασυνοριακές συνθήκες και που αφορά άμεσα όμως και την διεθνή κατάσταση και το κράτος δικαίου καθώς επίσης και το νομικό καθεστώς του λιμένος της τεριές της από τη στιγμή που πρόκειται για πλωτά ύδατα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μετά από απάντηση του Αυγούστου 2012 του Αρμοδίου Επιτρόπου πρέπει να πω ότι το ολιμένα της ε, ταιριές της ε, υφίσταται πλέον τις διαδικασίες και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 της συνθήκης, της συνθήκης Πάτσε. Ζώνη λοιπόν ελεύθερης ε, ναυσιπλοείας ε, διεθνούς ε, καθεστώτος. Επομένως το εσωτερικό των υδάτων του λιμένου στις τεριές της δεν ανήκουν μόνο στην Ιταλία και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστούν οι, τε, οι ιταλικές νομικές διαδικασίες οι οποίες απορρέουν και από, τις, ε, από την ε, ενωσιακή ε, νομοθεσία. Αυτές οι εγκαταστάσεις είτε οι της πανεριοποίησης είτε οι της offshore δεν συμμορφούνται λοιπόν με όλες αυτές τις διατάξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τζοραστάντε. από την Επιτροπή ο κύριος Κοντέσκου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτή η έρευνα διεξάγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε σε επαφή με τους αναφέροντες και γενικότερα οι ταιριέστοι είναι υπό πολλές έρευνες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω συνοπτικά για τα διάφορα ζητήματα και για τις εξελίξεις. Καταρχάς, τον, η νέα πιλωτική έρευνα που έχει σχέση με την εκαθάριση των SEA σε σχέση με τις τροποποιήσεις ε, που σχεδιάζονται για το λιμάνι της Τεργέστης και για τον χώρο εκφόρτωσης εκεί. Αυτά τα σχέδια δεν περικλείουν το εργοστάσιο επαναεριοποίησης, αλλά το λιμάνι. Αυτή η έρευνα συνεχίζεται. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τις Ιταλικές αρχές και φαίνεται πως ε, οι διαδικασίες, όπως από ό,τι γνωρίζουμε, έχουν τεθεί σε λειτουργία και για τα δύο σχέδια αυτά από τις Ιταλικές αρχές. Τώρα, κάτι σημαντικό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι Σύμφωνα με την οδηγία για τα SAA, για τις ΣΠΕ, το υποχρεωτικό είναι μόνο για τα υποχρεωτική έρευνα γίνεται μόνο για τα εργοστάσια που καλύπτονται. Και έτσι λοιπόν, για να, για να εναρμονιστούμε με αυτή την οδηγία, Σύμφωνα με την οδηγία για τα ΣΠΕ, ένα σχέδιο ή ένα πρόγραμμα πρέπει να ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Και καθώς φαίνεται, ούτε η Ευρωπαϊκή ούτε η Ιταλική νομοθεσία προβλέπουν κάποια υποχρέωση να υιοθετήσουν ένα ενεργειακό σχέδιο που να καλύπτει αυτά τα εργοστάσια επαναεριοποίηση. Και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή και η Ιταλική δεν είναι υποχρεωτικό να υιοθετηθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Όπως επίσης δεν είναι και υποχρεωτικό να υπάρχει μία ΣΠΕ για αυτά τα, σχέδια, τα εργοστάσια επαναεριοποίησης. Και όπως είπα και στην αρχή, οι Ιταλικές αρχές διεξάγουν στρατηγικές περιβαλλοντικές ε, μελέτες για το λιμάνι και για τα σχέδια για το λιμάνι της ταιριές της. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία σε Βέσο, είναι μια άλλη έρευνα που διεξάγεται έχει ολοκληρωθεί μία διαδικασία επιπαραβάση πέρυσι και αυτή η έρευνα είναι και πιο γενική, διότι αφορά και την εφαρμογή της οδηγίας σε Βέζο στην, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Τεριέστη, Όχι δηλαδή για το εργοστάσιο παναριοποίηση, διότι αυτά είναι σχέδια τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη. Υπάρχει μια νέα πιλωτική έρευνα επίσης που διεξάγεται σε σχέση με το άρθρο 6, δηλαδή το domino effect για όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην περιοχή. Μόλις λάβαμε ε, συμπληρωματικές απαντήσεις από τις Ιταλικές αρχές σχετικές με την αξιολόγηση και να τονίσω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό προς το παρόν δεν καλύπτει το εργοστάσιο παναεριοποίησης, δεν έχει χορηγηθεί έγκριση για αυτά τα εργοστάσια, έτσι, δεν καλύπτονται από τις ε, προδιαγραφές που υπάρχουν σε άλλες υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην Τεργέστη. Τώρα, για το εργοστάσιο πανεριοποίησης, που είναι η έρευνα που διεξάγουμε τον εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό. Έχουμε, όπως είπε και ο αναφέρον, τρεις εγκαταστάσεις. Αφορά τρεις εγκαταστάσεις και ενώ η κατάσταση από εγκατάσταση σε εγκατάσταση διαφέρει, θα σας τα πω σύντομα. Υπάρχει ένα μεγάλο ε, project στο Ζάουλε, το οποίο, στο οποίο, ε, για το οποίο μάλλον εκδόθηκε μία ΕΠΕ το 2003, αλλά δεν έχει χορηγηθεί καμία έγκριση. Και τι σημαίνει αυτό, δεν έχει εγκριθεί το σχέδιο ακόμα. Φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τις Ιταλικές αρχές, ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί έγκριση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον αγωγό φυσικού αερίου, το οποίο είναι το δεύτερο ε, σχέδιο στο οποίο θα αναφερθώ. Σύμφωνα με τις, σύμφων, με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις εξελίξεις, οι λιμενικές αρχές επίσης διεξάγουν αυτές τις ε, στρατηγικές περιβαλλοντικές ε, έρευνες και οι λιμανικές αρχές της Τεργέστης θεωρούν ότι προβλέπεται αύξηση στην ε, κίνηση στο λιμάνι και αυτό μπορεί να θέσει σε, να, να θέσει σε εμβολία στην ολοκλήρωση του τερματικού σταθμού. Μετά, σε συνέχεια αυτού, ο Ιταλός Υπουργός Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει μία νέα διαδικασία ΕΠΕ για το Ζάουλε και όπως είπα εκδόθηκε μια τέτοια αιτία το 2009, αλλά ενδέχεται να τροποποιηθεί από αυτήν την ε, επιπρόσθετη διαδικασία. Γι' αυτό το παρακολουθούμε στενά. Τώρα, το δεύτερο project, ο αγωγός φυσικού αερίου, που συνδέει αυτές τις onshore εγκαταστάσεις, που συνδέει δηλαδή και το, που συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου. Παρομοίως τώρα, δεν έχει δοθεί ε, έγκριση για την ανάπτυξη του έργου, και δεν έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία, η ερευνητική διαδικασία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης πληροφορήθηκε ότι η Σλοβενία ενημερώθηκε, αλλά η διαδικασία ΕΠΕ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το τρίτο project είναι το offshore project στη θάλασσα και έχουμε και εδώ παρόμοια περίπτωση. Δεν έχει χορηγηθεί ακόμα έγκριση, δεν έχει ολοκληρωθεί η ΕΠΕ. Και σύμφωνα με την ε, θέση των λιμενικών αρχών της Τεριέστης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αρχίσει περαιτέρω έρευνες σε συνδυασμό με την, και παράλληλα με την ε, ΕΠΕ. Και στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται μπορεί να λάβουν υπόψη του τις ανησυχίες που διατύπωσε ο αναφέρον. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Ιταλικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι αυτό αφορά και άλλα κράτη-μέλη και την Κροατία και πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις και να κρατούνται όλοι ενήμεροι από τις Ιταλικές αρχές. Και κάτι που θα ήθελα να τονίσω κλείνοντας, είναι το εξής. Όπως αναφέρθηκε και από τους αναφέροντες, αυτά τα project δεν έχουν εγκριθεί και έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθούμε σε κάποιο τελικό και οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το πώς οι ε, προϋποθέσεις για τις ΕΠΕ καταρτώνται και πώς διεξάγονται οι ΕΠΕ. Η τελική συγκατάθεση για τα project αυτά με το φυσικό αέριο θα μας δώσουν την ευκαιρία να δούμε πώς ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί η οδηγία για τα ΕΠΕ και, πώς, και πού θα μας οδηγήσουν οι δημόσιες διαβουλεύσεις. Φυσικά στο μεταξύ έχουμε αξιολογήσει όλες τις πληροφορίες που λάβαμε από τους αναφέροντες, από τις Ιταλικές αρχές. Υποβα... Υποβάλλουμε τακτικά ερωτήσεις στις Ιταλικές αρχές και ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις. Όμως η οδηγία για τις ΕΠΕ, όπως συζητήθηκε και σήμερα το πρωί, ε, ρέχει κάποιο πλαίσιο σε ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σύμφωνα με την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μόνο όταν υπάρχουν λάθη στην... στις ε, ΕΠΕ και όχι συγκεντρωτικά, ε, για παράδειγμα μάλλον συγκεντρωτικές επιπτώσεις, τότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε και να διεξάγουμε <clears throat> τις έρευνες. Μέχρι όμως τώρα δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας και από ό,τι καταλαβαίνω και σύμφωνα με, την, με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν έχουμε εντοπίσει λοιπόν τέτοια οφθαλμοφανή λάθη. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να αποδείξει ότι υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των ε, πληροφοριών που είχαμε για να κάνουμε την αξιολόγηση. Όπως είπαμε και στην ε, ανακοίνωση, χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για να εντοπίσουμε λάθη και παραβιάσεις. πέρα από κάθε αμφιβολία, να είμαστε σίγουροι προτού ξεκινήσουμε διαδικασία επί παραβάση. Και όπως είπα δεν έχει εντοπιστεί κάποια παραβίαση μέχρι τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε ακόμα την τελική έγκριση για την ε, ανάπτυξη σύμφωνα με την, ε, με την οδηγία περί συντονισμού. Για παράδειγμα, ε, οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να δείξουν με τη συγκατάθεσή τους τα αποτελέσματα της, ε, των διαβουλεύσεων. Και τώρα, όσον αφορά τον, ε, την ποιότητα του αέρα, το τελευταίο σχόλιο, η Ιταλία από τον Νοέμβριο, το Δεκέμβρη πέρυσι, έχει θέσει κάποια πρότυπα για την ποιότητα του αέρα και αυτό λόγω των ε, βιομηχανικών εκπομπών. Και αυτό το έχουμε λάβει υπόψη και καθώς γνωρίζετε φέτος είναι η χρονιά για την ποιότητα του αέρα και διεξάγονται προς το παρόν διάφορες ε, διαδικασίες παραβάση για πολλά κράτη-μέλη και παρακαλουθούμε τις εξελίξεις σε αυτό και έχουμε ζητήσει από τις εθνικές αρχές να επιληφθούν του θέματος. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ εγώ πολύ. Ήταν πολύ αναλυτική η παρουσίαση. Ε, να προχωρήσουμε. Ο κύριος Κλέβα, ε, η κυρία Κλέβα ζήτησε την, να μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Μόνιτσα Κλέβα. Από το δίγλωσο... Ε, ε, περιβάλλον της ε, Ίστρια. Είμαι όμως εκλεγμένη ως Σλοβαίνη βουλευτήνα. Αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις είναι δύσκολες. Εγώ ζω, ζω σε αυτόν τον κόλπο της ταιριές της στην ουσία και με ενδιαφέρει άμεσα σαν ε, πολίτη της ε, ε, Σλοβενίας η εξέλιξη αυτών των δύο εγκαταστάσεων. Κατά την άποψή μου, η παρέμβαση του εκπροσώπου της Green Action και της σλοβενικής πλευράς σε αυτήν την αναφορά της Alpe Adria Green ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, λέω, οι παρεμβάσεις αυτές. Ε, γιατί αυτό το θέμα της ε, επανεριοποίησης είναι hot topic, είναι καυτό ζήτημα. Και σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε ακόμα περισσότερο βέβαια, σε τοπικό επίπεδο. Στην Ιταλία και στην Κροατία είδαμε όμως ότι ο κόσμος δεν είχε την δυνατότητα ε, να εκφράσει την άποψή του όσον αφορά είτε εναλλακτικέ ε, περιοχές εγκατάστασης, είτε και για την ίδια την ε, επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων αυτών. Ελπίζω ότι μια και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Κυρίω Κυρίως όσον αφορά το θέμα της ε, πλαστογράφησης ε, ε, τη της, περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Gas Natural, όπου φαίνεται ότι απεκρίβησαν οι μεγάλοι κίνδυνοι για το περιβάλλον, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο κατά την άποψή μου. Και βεβαίω οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται μονάχα ε, στο περιβάλλον. Δηλαδή έχουμε γεωλογικού κινδύνους, περιβαλλοντικού κινδύνους, κινδύνους μόλυνσης των ε, υδάτων, κινδύνους παρακόλλησης ε, των θαλασσίων μεταφορών κλπ. ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ήταν σαφής και μας εξήγησε σε αρκετή λεπτομέρεια πώς βλέπει την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, εγώ έχω μία αμφιβολία όσον αφορά το, την κατάθμιση ε, του σχεδίου σε δύο τμήματα. Ε, εντάξει, ε, αυτό το πρώτο κομμάτι της Gas Natural, ας πούμε το καταλαβαίνω, αλλά αυτός ο, ο αγωγός ε, διασύνδεσης με το Εθνικό Δίκτυο Αερίου με προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Ε, ε, νομίζω ότι αυτή είναι μια κατάτμιση η οποία ε, είχε σαν μόνο κίνητρο την υποβάθμιση της σημασίας της ΕΠΕ και την ανάγκη ύπαρξης ΕΠΕ και στρατηγικής αξιολόγησης. Θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα από κοντά. Και θα πρέπει βέβαια να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά ε, στοιχεία, γιατί πολλά διαβάζουμε και στον τύπο, στο δικό μας τύπο τουλάχιστον, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε όλα τα στοιχεία. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο ούτε ένας πια δεν πιστεύει σε αυτό το ε, σχέδιο. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δήμοι και αυτός από τον οποίο προέρχομαι εγώ αλλά και ε, άλλοι αποφάσισαν ε, να δώσουν αρνητική γνωμοδότηση, πράγμα όχι πολύ συνηθισμένο στα δικά μας τα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των ευρωπαϊκών συνθήκων ίσως θα πρέπει να ξαναδεί το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από τη Σλοβενία. Θα ήθελα να τονίσω όμως ότι αυτός ο τερματικός σταθμός δεν είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα για τον ε, τοπικό πληθυσμό, όχι μόνο για το κοινό της Σλοβενίας, αλλά το να ξανανοίξουμε την ε, ενεργειακή έκθεση του Ιταλού Υπουργού Περιβάλλοντος είναι κάτι το αυτονόητο. Ο κύριος Τζιραστάντε και η κυρία Σκλέιβα μας εξήγησαν ακριβώς πώς γίνεται η διαδικασία εφοδιαστικής, ποιες ανησυχίες υπάρχουν για την ασφάλεια. Θα ήθελα εγώ όμως να πω ότι το θέμα δεν είναι μόνο διαδικαστικό και διοικητικό, αλλά υπάρχουν υπαρκτοί περιβαλλοντικοί προβληματισμοί, υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Πιστεύω πως είναι το σοβαρότερο. Η ύπαρξη υδράργυρου στο βόρειο τμήμα της Αδριατικής. Ο υδράργυρος αυτός ε, εναποτίθεται για αρκετούς αιώνες στο βόρειο τμήμα της ε, θάλασσας εξαιτίας των ορυχείων στην ίδρια υδράργυρου. Τώρα λοιπόν υπάρχει υδράργυρος εκεί αλλά εξαιτία των δραστηριοτήτων ο βυθό τη θάλασσα θα διαταραχτεί και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για αύξηση των ε, επιπέδων του υδράργυρου και για ανάμειξή του και για διάχυσή του στο οικοσύστημα και σε άλλα μέρη. Υπάρχουν λοιπόν σοβαροί προβληματισμοί για το περιβάλλον. Τώρα όσον αφορά την ενεργειακή ε, παροχή και την ασφάλεια υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα Ξέρουμε πλέον ότι το South Stream συνεχίζεται, έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς ε, την ολοκλήρωσή του. Επίσης υπάρχει το, ε, το εργοστάσιο στο Ναμπούκο και αυτοί οι δύο τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν είναι πλέον στην πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω κλείνοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, η Σλοβενία να διατυπώσει ε, νομική, νομικό παράπονο μετά την κατασκευή των δύο αυτών τερματικών σταθμών. Η Σλοβενία θα πρέπει να περιμένει για την τελική έγκριση έτσι ώστε να διατυπώσει δικαστικά τις αντιρρήσεις της. Θα ήθελα λοιπόν να το αποτρέψουμε αυτό. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που συνεισφέρατε σε αυτή τη συζήτηση. Όσοι δεν γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό το έργο. Μήπως όμως το 2008 είχαμε συζητήσει κάτι πολύ παρόμοιο που είχε να κάνει με το North Stream. Τώρα βέβαια σε μικρότερη κλίμακα μεν, αλλά είναι ένα είδος North Stream. Στην Αδριατική αυτή τη φορά. Πρώτον, εδώ έχουμε το ζήτημα της διασυνοριακής διάστασης αυτού του project. Και η Κομισιόν προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα για τη, με την τροποποιημένη πρότασή της για τη ΣΕΠΕ. Και βέβαια, φυσικά, το project αυτό δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Λοιπόν, που το λέω αυτό, αλλά η Ιταλία δεν μπορεί να επιβάλλει το project αυτό ενάντια στην βούληση, αλλά και τις νομικές αρμοδιότητες και ξέρεις, της Σλοβενίας και της Κροατίας. Και ιδίως από πλευράς διεθνούς δικαίου λόγω της πόλης ταιριές της και του λιμανιού της. Θα πρέπει εκ των προτέρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ΕΠΕΙΣΠΕ αν δεν έχουν πρώτα επιληθεί τα νομικά ζητήματα. Γιατί πώς μπορεί κανείς να επιβάλλει μια ΕΠΕ σε ένα φορέα, σε μια οντότητα που αναγνωρίζεται ως διεθνής φορέας. Ήταν υποχρεωτικό κάθε κράτος <clears throat> μέλος το οποίο άμεσα συμμετείχε στο Nord Stream ή και όχι να αποδεχθεί νομίμως την ΕΠΕ. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο εδώ, τουλάχιστον δεν μας είπε η Κομισιόν ότι δεν μπορεί να γίνει ΕΠΕ και να θεωρηθεί έγκυρη αν πρώτα δεν έχει ρητά γίνει αποδεκτό αυτό από όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, μεταξύ αυτών και από τη Σλοβενία. Δεύτερον, έχοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του project και από νομικής πλευράς και από περιβαλλοντικής πλευράς, είναι πολύ σημαντικό να δει κανείς και την ε, ΣΠΕ αλλά και την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πρέπει να δούμε γιατί μιλάμε πιο πολύ για ΕΣΠΕ ή για ΕΠΕ. Και θα πρέπει εκ των προτέρων αυτό να το έχουμε εξετάσει και να έχουμε καταλήξει. Μπορεί κάτι να κάνει η Κομισιόν λοιπόν για να καταρτήσει ένα πλαίσιο για ένα τόσο πολύπλοκο project και για τη μελέτη και το σχεδιασμό του αφενός και για την αποδοχή του και ε, την εφαρμογή του αφετέρου. Αν δεν ολοκληρωθούν αυτά τα προκαταρκτικά στάδια από την Κομισιόν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλιώς θα φτάσουμε να πούμε, ναι, μοιραία έγινε, τι να κάνουμε. Επίσης, δεν υπάρχει μνήα στα προβλήματα ασφάλειας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αντιμετωπίσει τους ενδεχόμενους τρομοκρατικούς κινδύνους που σχετίζονται με ένα τέτοιο project. Οι Ιταλοί θα είναι οι Σλοβαίνοι, θα είναι κοινέ δυνάμεις, θα είναι το ΝΑΤΟ, θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αναλάβει αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι κενό. Στην περίπτωση του Nord Stream, ποιος θα πάρει την έγκριση, για παράδειγμα, για εισόδηση στα εθνικά έδατα. Είναι ζήτημα ασφάλεια. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τι στρατιωτικά μέσα, τι τεχνικά μέσα απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων ή η αξιολόγηση κινδύνων, το ενδεχόμενο καταστροφής, όπως είχαμε στον κόλπο του Μεξικού. Ποιο θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με τι τεχνικά μέσα. Και τέλος, ούτε μία λέξη δεν ακούσαμε ή διαβάσαμε για τα νομικά εχέγγυα και για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια καταστροφή. Η εταιρεία, ο επενδυτής αυτός, έχει την ικανότητα, έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να καλύψει όλες τις οικονομικές και νομικές αποζημιώσεις σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Ούτε μια λέξη δεν έχει λεχθεί γι' αυτό. Τώρα, Καλός ή κακός, ο Επίτροπος Αρμόδιος για το Περιβάλλον είναι από τη Σλοβενία. Και ως Ποτότσινικ ελπίζουμε, στην αυτή η περίπτωση τουλάχιστον, να αντιμετωπίσει και τα δυσυνοριακά προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και η Κομισιόν να μπορεί να έχει έναν λόγο νομικά δεσμευτικό για τα θέματα αυτά. Αλλιώς το μόνο που θα γίνει θα είναι ότι δεν θα έχουμε κανένα περιθώριο ούτε να πούμε ούτε να κάνουμε τίποτα εμείς. Και οι παντοδύναμες οικονομικές δεσμεύσεις θα υπερισχύουν, θα υπερτερούν έναντι των συμφερόντων ορισμένων κρατών μελών. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει τα απαραίτητα νομικά εφόδια για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Η πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποστίνα. Ο Μποστίνα. Ναι, πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Η πρόεδρο, ναι, φυσικά και θα παραμείνει ανοιχτή. Και νομίζω ότι πράγματι υπάρχει εδώ ένα νομικό κενό που δείχνει και την ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι χώρε δεν είναι απλά ε, κρατημέλη, είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα η Κομισιόν πρέπει κάτι να κάνει σε αυτό το μέτωπο. Από ό,τι έμαθα, υπάρχουν επιστολές και προς την Ιταλική και προς την Σλοβενική κυβέρνηση. Ο κ. Ποστινάρ, με συγχωρείτε, η Κροατία δεν είναι μεν επισήμως ακόμη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από νομικής πλευράς η Κροατία έχει υπογράψει. Έχει υπογράψει και έχει επικυρώσει όλες τις νομικές πτυχές που άπτονται της ε, κατάστασης ε, κράτους μέλους. Στην ομολογία προβλέπεται ότι όπου άπαξ και εγκριθούν και επικυρωθούν οι νόμοι, παράγουν να έχουν νομικές επιπτώσεις. Επομένως και η Κροατία θα πρέπει να αποτελέσει παραλήπτη της αλληλογραφίας, της σχετικής. Αν η Κροατία δηλαδή συμμετάσχει σε αυτό το project και δεχθεί, θα πρέπει να αναλάβει και να φέρει σε πέρας και τις δικές της ευθύνες και υποχρεώσει. υποχρεώσεις. Πρόεδρος, άρα συμφωνείτε να σταλούν επιστολές στι κυβερνήσει, επομένω, Ιταλίας, Σλοβενία και Κροατίας. Και βέβαια παραμένει ανοιχτό το θέμα. Έκλεισε το μικρόφωνο του Προέδρου. Uh, petition number 18. λοιπόν στον κύριο Διάννα. Ε, για την αναφορά 18. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε το έγκριτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δέχτηκε την αναφορά μας και που μας έδωσε τη δυνατότητα να τη συζητήσουμε εδώ όλοι μαζί. Στην αναφορά αυτή διαμαρτυρόμεθα, ε, καταγγέλουμε την απόφαση ε, για χρηματοδότηση της εγκάλση με 120 εκατομμύρια ε, ευρωπαϊκών πόρων και αναφερόμαστε στον οργανισμό 663-2009 και τις ακόλουθες τροποποιήσεις τους. Ε, βρισκόμαστε εδώ διότι οι ε, προϋποθέσεις δεν έχουν ε, καλυφθεί και επίσης και οι απαντήσεις που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν σε θέση να να απαντήσουν πραγματικά στις ερωτήσεις μας όσον αφορά την συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά την κάλυψη που ευτυχώς σαφώς τώρα πλέον δεν είναι από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς αναφερόμαστε ε, και σε κάποια ζητήματα τα οποία αμφισβητούμε όσον αφορά την κάλυψη. Πρώτον, το βαθμό οριμότητας του ε, σχεδίου ε, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Νόμο και που θα πρέπει η οριμότητα αυτή να θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 2010. Όσον αφορά την επίπτωση του σχεδίου επίσης αμφισβητούμε το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη περιβαλλοντική, ε, ε, ε, πολιτιστική και άλλοι όροι. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δεν έχουν ε, τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης, ασάφεια ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Και πέμπτο σημείο, η αναξιοπιστία του σχεδίου όσον αφορά την εταιρική σχέση που ε, έχει προβλήματα, όπως γνωρίζουμε, με την δικαιοσύνη και όσον αφορά την έλλειψη απόφασης παρέμβασης, καθώς επίσης και την έλλειψη οποιασδήποτε προγραμματικής εθνικής, ε, ε, εθνικού συγγνώμη, ή περιφερειακού προγραμματισμού. Ε, όσον αφορά την οριμότητα του σχεδίου, την οποία να αμφισβητούμε και η οποία όμως απαιτείται από τον νόμο. Αναρωτιόμαστε πόσο όριμο μπορεί να είναι ένα σχέδιο ε, προμήθειας αερίου χωρίς αέριο. Η Αλγερία, από όσο γνωρίζουμε, δεν προτίθεται να πωλήσει το αέριο ε, στους, ε, υπό τις παρούσες συνθήκες και δεν ξέρουμε πότε θα αλλάξει γνώμη. Επομένως δεν υπάρχει πρώτη ύλη να μεταφερθεί. Και εδώ μπορώ να σας ε, παραπέμψω στις ε, δηλώσεις τις οποίες έκαναν οι σύμβουλοι της Αργυρινής Κυβερνήσεως ε, σε ένα φιλμ έρευνας που, γύρισε, που γύρισαν κορσικανοί δημοσιογράφοι που ενδιαφέρονται και αυτοί ως προερχόμενοι από την Κορσική της, του τρίτου προγράμματος γαλλικής τηλεόρασης και που ονομάζεται «Προπέτασμα καπνού», εκράνονται Εφημέ. Όσον αφορά το περιβάλλον τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Γκάλση θα έπαιρνε αυτήν την περιφερλοντική ε, αδειοδότηση σε σχέση με την ΕΠΕ. Όμως τίποτα δεν έχει γίνει. Η μόνη αδειοδότηση που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η οποία σχετίζεται με την ε, ε, κατασκευή του αγωγού. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία ΕΠΕ. Ε, η ΕΠΕ μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν επιτρέπει τίποτα. Ε, αντιθέτως μάλιστα επιβάλλει 112 δεσμευτικές προδιαγραφές με καμία δε από τις οποίες ε, δεν υπάρχει συμμόρφωση. Ε, και επίσης το ίδιο συμβαίνει και με την, ε, με την απόφαση 357 του 97 που δεν ζητήθηκε ποτέ ε, η συμμόρφωσή της από τις Ιταλικές αρχές. Εξακολουθεί πάντως να υπάρχει πολύ αρνητική επίπτωση στα περιβάλλοντα ε, οικοσυστήματα. Έχουμε, ας πούμε, το, ε, την, το, το ωκεανικό ε, οικοσύστημα της Ποσειδόνια, που θα έπρεπε να επιβάλλει τροποποίηση της, του περάσματος αυτού του αγωγού. Γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη απικία πίνα νόμπιλης στην Μεσόγειο και αυτό φαίνεται αν το όλοι. Επίσης, ε, ε, όσον αφορά το, ε, την αδειοδότηση τη βάση της ΕΠΕ σχετικά με το κέντρο συμπίωσης, συμπίκνωσης της Όλμπια και εκεί δεν είναι δυνατόν να δοθεί μια τέτοια αδειοδότηση. Επίσης, ε, ξέρουμε ότι περνάει από πολύ σημαντικά, ε, ε, από πολύ σημαντικά οικοσυστήματα ο αγωγός αυτός. Επίσης, αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνονται υπόψη είναι και όλα τα υπόλοιπα αρχαιολογικά ευρήματα γιατί στην περιοχή αυτή δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε 8 νουράγγι αυτά τα προϊστορικά κτίσματα της εποχής του Χαλκού που οπωσδήποτε θα πρέπει ε, να καταστραφούν εάν περάσει από εκεί το σχέδιο. Ε, στο εκράνο του αυτό το φιλμάκι στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, ε, βεβαίως όλα αυτά αναφέρονται μαζί και με την εκρίζωση των αμπελώνων και τον, την, την πάυση των δραστηριοτήτων αγροτουρισμού κτλ. Όλα αυτά αναφέρονται λοιπόν. Επομένως ε, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία αντιτίθενται ε, στον προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το 2020. Επομένως πιστεύουμε ότι οι μόνοι που πιστεύουν στην ορθότητα του προγράμματος είναι ε, οι εταιρείε. Όμως πρέπει να πούμε ότι έπρεπε να είχαν υπογράψει μέχρι το τέλος του 2010 οι εμπλεκόμενες εταιρείε και αυτή την απόφαση επένδυσης ε, σύμφωνα με, τον, ε, ε, Ευρωπαϊκό, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τέτοια υπογραφή δεν έχουμε δει. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα και την αναξιοπιστία του προγράμματος, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ασάφεια όσον αφορά την θέση σε εφαρμογή. Μάλιστα η αρχική θέση ισχύει προβλέπεται για το 2009, φανταστείτε λοιπόν. Επίσης δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα προγραμματικά ε, ε, σχέδια είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο και καμία ανάλυση κόστους οφέλους. Ε, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γκάλση θα περάσει ένα από τα πιο παλαιά αρχαία νησιά της Ευρώπης ε, που έχει δάση, που έχει ελαιώνες, που έχει αμπελώνες, που έχει αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που έχει ε, προστατευμένες περιοχές κτλ. Ποτάμια, λίμνες και αυτά. Οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε ότι είναι τεράστιες οι επιπτώσεις που θα είχε στο περιβάλλον, στο πληθυσμό και στην ε, κοινωνία. Επίσης, δεν υπάρχουν υδρογεολογικοί και αρχαιολογικοί χάρτες. Για να μην αναφέρω το γεγονός ότι και η Σόνατρακ και η Ένη ε, ελέγχονται για διεθνή διαφθορά από την εισαγγελία του Μιλάνου. Ε, οι συναντήσεις κορυφής της Σόνατρακ διαρκώς αναβάλλονται λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων με την δικαιοσύνη. Ε, και ε, δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι προσφάτως διαβάζουμε και στον αλγερινό τύπο και πολύ σημαντικές τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του αερίου. Συμπερασματικά μπορώ να πω ότι εδώ μιλάμε για ένα από αυτά τα μεγάλα άχρηστα έργα, τα οποία πολύ σωστά αναλύει ο γνωστός ε, γερμανός ε, οικονομολόγος Βίλφιντ Βόλφ. Ε, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μιλάμε για ένα τέτοιο σχέδιο, γιατί η γκάλση δεν έχει συμμορφωθεί καθόλου με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν έχει όριμο σχέδιο, δεν έχει καμία πρόβλεψη όσον αφορά την τρομακτική καταστροφή στο περιβάλλον στην οικονομία, στην κοινωνία. Ε, δεν ε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν συμμορφώνεται καθόλου, δεν, ε, ευθυγραμμίζεται καθόλου μάλλον με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές κλπ πρέπει να σας πω ότι ε, εμείς θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι από τη στιγμή ε, που ε, έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία στην διάθεσή μας, έχουμε σκοπό να προστρέξουμε και να προσφύγουμε σε, όλες τις, σε όλους τους φορείς στους οποίους μας δίνεται η δυνατότητα να προσφύγουμε και εκπροσωπούμε όλους τους κατοίκους του νησιού μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διάννα. παρακαλώ από την Επιτροπή κυρία Εζινάρ. Merci Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω. Είναι ίσως σημαντικό να υπενθυμίσω το πλαίσιο. Αυτό λοιπόν το project εντάσσεται σε project επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος ε, βοήθειας για την ανάκαμψη. Το εγκρίναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αυτό το πρόγραμμα, οπότε επελέγησαν ε, σε βέβαια καιρού οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ορισμένα project το 2009-2010. Είχαμε βέβαια κρίση και στο τομέα του φυσικού αερίου και επελέξαν αυτά τα project για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εφοδιασμού της Ένωσης σε φυσικό αέριο. Αυτά λοιπόν τα project συνολικά πρόκειται για έργα υποδομών για παροχή ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και επελέγησαν γιατί θεωρούσαμε ότι συμβάλλουν στους στόχους ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών, δηλαδή την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ε, το να πάψουν να υπάρχουν ενεργειακές νησίδες Συγκεκριμένα ο εν λόγω αερογός μέσω Σαρδινίας εφοδιάζει την Ιταλία και μπορεί να φτάσει μέσω Κορσικής και στην Γαλλία, ε, ουσιαστικά δηλαδή να εφοδιάζει την Κορσική. Η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτό το έργο έχει και σημαντικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, διότι παρέχει ουσιαστικά ένα νέο, μια νέα διαδρομή για το αέριο από την Αλγερία μέσω Ιταλίας. Θα μπορούσαν ενδεχομένω να εφοδιαστούν και άλλα κράτη-μέλη, τα κράτη δηλαδή ε, βόρεια και ανατολικά και δυτικά μάλλον της Ευρώπης, επίσης, της Ιταλίας. Επίσης θα μπορούσε να υπάρχει και διαφοροποίηση των προμηθευτών, γιατί με αυτό το έργο μπορεί το φυσικό έργο να από την Ιταλία με κοινοπραξία που έχουμε τη Ωνατρακ, αλλά και οι Ιταλικές, την Edison και την Eni, και στη Σαρδινία συμμετέχει η εταιρεία αυτή της Σαρδινίας, άρα και η περιφέρεια της Σαρδινίας εκπροσωπείται. Άρα θεωρούσαμε στρατηγικό αυτό το project στο πλαίσιο ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και γιατί εντάσσεται στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, αλλά και γιατί θεωρείται ένα project οικονομικού ενδιαφέροντος εξού και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ανάπτυξη, την ε, εξέλιξη αυτού του έργου, ξέρουμε ότι είναι στη φάση ε, της, εξέλιξης εξέλιξη είχαμε τις περιβαλλικές ε, μελέτες το 2011. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και η Ιταλία θα πρέπει να εξηγήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποιο τρόπο έλαβαν υπόψη ε, κατά την κατασκευή του έργου τις διάφορες παραμέτρους που να κάνουν με την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη των έργων, είναι σε εξέλιξη διοικητικές διαδικασίες, στην τελική φάση, άρα περιμένουμε τις εγκρίσεις, τις διοικητικές εγκρίσεις για να μπορέσει να αρχίσει κατασκευή στο πρώτο τρίμηνο ή εξάμηνο του 2013. Τώρα προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν προχωρήσει δηλαδή παραγγελία αγωγών φυσικοαερίου, σωλήνων, γιατί χρειάζεται χρόνος για την παραγγελία. Από τεχνική πλευρά είναι πολύπλοκο δηλαδή το όλο project. Ε, υπάρχουν ε, προκατακτικέ εργασίε που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και μετά να ξεκινήσει ουσιαστικά ε, η κατασκευή του έργου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, μέχρι στιγμής η απόφαση για την επένδυση δεν έχει ληφθεί ακόμη για μεγάλα έργα υποδομών που, στα οποία συμμετέχουν διάφορα άρα υπάρχουν και διάφοροι εταίροι, περισσότεροι του ενός και βέβαια τα ποσά είναι πολύ ψηλά. πάνω, είμαστε πάνω από το ένα δις για, για το συγκεκριμένο project. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι συμμετέχοντες, εμπλεκόμενοι και καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται χρόνος και η απόφαση για να ε, υπάρξει επένδυση δεν λαμβάνεται εύκολα και αβασάνιστα. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση, δόθηκαν τα κονδύλια, ε, ανατέθηκαν, αλλά η εκταμείευσή τους θα γίνει μόνο αν έχει πάρει περιβαλλοντική έγκριση το project και αν διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται σωστά και τηρούνται οι υποχρεώσεις. Δηλαδή, Πρόσταση ορισμένων ειδών, ό,τι περιλαμβάνεται τέλο πάντων στην ε, περιβαλλοντική έγκριση. Και έπειτα η εκταμείευση θα γίνει όταν ο εργολάβος θα καταδείξει ότι υπήρξε και απόφαση για επένδυση, για τις επενδύσεις που χρειάζονται. Ναι. Ε, περιμένουμε με αγωνία την εκτίμηση για τις περιβαντολογικές επιπτώσεις από τη μεριά της Κομισιόν, ομολογουμένως, γιατί από όσα ακούσαμε από την ε, Σαρδινία υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και όχι μόνο περιβάλλοντος και αρχαιολογικού και πολιτικής κληρονομιάς και τέτοια. Ελπίζω ότι θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη πριν ξεκινήσει η χρηματοδότηση αυτού του τεράστιου έργου. Επομένως προτείνω, αν δεν έχει αντίρρηση κανείς, να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, ε, υπόθεση, την αναφορά, περιμένοντας με αγωνία θα έλεγα και πριν από τη χρηματοδότηση, ε, την έγκριση της χρηματοδότησης, της, ε, την ΕΠΕ, της, τη μελέτη περιβαλλοντολογικών και άλλων επιπτώσεων. Και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση προκειμένου να μην καταστραφεί τίποτα από αυτά για τα οποία μας μίλησε ο κύριος Διάννα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε. προχωρούμε στην επόμενη. Ε, πάμε στην Ιρλανδία από τη Σαρδινία τώρα για ένα θέμα παρόμοιο με υγροποίηση φυσικού αερίου. Παρακαλώ τον ε, κύριο Έλγκοτ να παρουσιάσει την αναφορά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα εδώ. Έχουμε δύο ζητήματα που μας ανησυχούν για το project του ποταμού Σάνων. Καταρχάς δεν έγινε καμία ΣΠΕ και καμία μελέτη θαλάσσιου κινδύνου. Για το πρώτο θέμα, για την έλλειψη δηλαδή ΣΠΕ, τα άρθρα 1 και 3 της οδηγίας για τη ΣΠΕ απαιτούν να διεξαχθεί ΕΠΕ για σχέδια τα οποία ενδέχεται να έχουν έστω και ελαφρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υπάρχει ένα πλαίσιο ανάπτυξης και συγκατάθεσης για τέτοια έργα, όπως για παράδειγμα τερματικού σταθμού συγκροπημένου φυσικού αερίου. Τι γίνεται εδώ πέρα. Το project για το Σάνον ψηφίστηκε το 2006 από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Δαπανήθηκαν περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ για την γη που αγοράστηκε και αυτό το project είναι ένα project που οποιοδήποτε ουδέτερος παρατηρητής θα έλεγε ότι εντάξει θα, διεκπε... θα ε, διεκπεραιωθεί. Όμως, στο στάδιο της ανάπτυξης δεν, ε, δεν μπορούσε, είχε μείνει στο στάδιο της ανάπτυξης μέχρι η αγροτική περιοχή να ε, άλλαζε και να γινόταν, σε, ε, να γινόταν πόλεο δομική περιοχή η διατύπωση το Μάρτιο του 2007 για την αλλαγή αυτή στην πολυοδομική ζώνη δεν έγινε ποτέ. Ε, τώρα σας καλώ να κοιτάξετε το άρθρο 1 και τη διατύπωση και να μου, και να μου πείτε εάν οι συνέπειες για την ε, επανονομασία της ε, ζώνης περιλαμβάνονται. Έγινε ένα σχέδιο στρατηγικού σχεδίου για, το, για τις εκβολές του Σάνων και έχει εκδοθεί τώρα και πιστεύουμε αυτό έγινε χάρη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την εποπτεία της. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό είναι περιορισμένο, διότι δεν μπορεί να εκτιμήσει εναλλακτικέ λύσεις για το έργο αυτό, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην Ιρλανδία είναι η μόλυνση του των εκβολών του ποταμού Σάνων και αυτό έχει ξεφύγει και δεν έχει γίνει όπως προβλεπόταν. Τώρα, στο δεύτερο ζήτημα, στην έλλειψη δηλαδή μιας εκτίμησης σε θαλάσσιο κινδύνου, οι Ιρλανδικές αρχές δήλωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν συμβουλευτεί επαρκώς από την HSA, δηλαδή την Ιρλανδική ε, Αρμόδια Αρχή ε, Υγείας και Ασφάλειας, για τις θαλάσσιες απόψεις του ε, Project Shannon. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτα διότι οι συμβουλές αυτές ήταν μόνο εκείνες που είχαν σχέση με την ε, περίπτωση όπου ένα πλοίο της εταιρείας αυτής ε, αγκυροβολούσε στο, ε, στον χώρο αυτό και αυτό δεν αφορούσε τους κινδύνους που προέκυπταν από τα, τα πλοία που ταξίδευαν στα νερά των εκβολών. Έχω υποβάλει επίσης ε, αποδεικτικά στοιχεία για αυτό και σας ζητώ να τα αξιολογήσετε. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει ήδη ασχοληθεί με μια πολύ ε, όμοια αναφορά για του δύο τερματικού σταθμού στο Milford Haven και στις εκβολές του Κλεντάου στην Ουαλία. Ζητώ να εφαρμοστεί το προηγούμενο που δημιουργήθηκε από τις αναφορές 4 του 2006 για το Milford Haven και το Κλεντάου. Επίσης, σημειώστε ότι διαφορετικά από ότι το Milford Haven, το project για τον ποταμό Σάνων δεν έχει αρχίσει ακόμα, οπότε έχετε αρκετό χρόνο. Και χωρίς μία εκτίμηση θαλάσσιου κινδύνου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ε, επιπτώσεις στην ασφάλεια, στο περιβάλλον και τις ε, σορευτικές επιπτώσεις που θα έχει η κίνηση και οι ζώνες αποκλεισμού στο δέλτα του ε, ποταμού Σάνων μέχρι ότου ολοκληρωθεί το project. Και αυτό θα σταματήσει το, τις εκβολές του ποταμού Σάνων ε, από το να εκπληρώσουν όλες τους ε, τις δυνατότητες. Και η αρμόδια αρχή έχει ήδη δηλώσει ότι το πόρισμα που θα δώσει αποκλείει οποιαδήποτε εκτίμηση άλλων ε, τύπων εγκαταστάσεων, λιμενικών εγκαταστάσεων, εκτός από τον τερματικό σταθμό. Εμείς πιστεύουμε ότι οι Ιρλανδικές πολιοδομικές αρχές δεν πρέπει να ε, μπορέσουν, δεν πρέπει να γνωρίσουν ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα του Ευρωπαϊκού Νόμου, τον οποίο άλλωστε έχουν υπογράψει και εγκρίνει. Βρίσκομαι στη διάθεσή σας, σας ζητώ να κρατήσετε την ε, αναφορά μου ανοιχτή και ε, είμαι στη διάθεσή σας για περιττέρω πληροφορίες. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και στην εθνική νομοθεσία και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, στην Ουαλία και στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ. From the commission από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Πέιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα να ακούσω απευθείας ε, τον αναφέροντα που όπως καταλαβαίνετε για πολύ καιρό έχει προετοιμάσει ε, την ε, παρουσίασή του τα θέματα τα οποία έθεσε που έχουν να κάνουν με την οδηγία ΕΠΕ, την οδηγία με τους οικοτόπους ε, και την οδηγία σε βέσο. Εμείς από την πλευρά μας ε, για να εξετάσουμε στην ουσία την αναφορά χρειάστηκε να ξεκινήσουμε διαδικασία pilot με τις ελληνικές Αρχές. Συναντηθήκαμε και μαζί τους, συζητήσαμε τα θέματα που θίγει ο αναφέρον και ξεκινήσαμε και μια διαδικασία επί παραβάση για ε, θέμα που ήταν σχετικό βέβαια, όχι άμεση απόρρια της αναφοράς. Ε, θα ήθελα να απαντήσω για τα δύο ζητήματα που θέτει σήμερα ο αναφέρον. Σας ευχαριστώ γιατί ήδη από χθε ε, μας στείλατε την εισαγωγική σας ομιλία που μας βοήθησε πάρα πολύ. Έλλειψη λοιπόν ε, ή μη διεξαγωγή ΣΠΕ για, τις για τα περισσότερα σχέδια χρήσης γης, όταν δηλαδή χρειάζεται και ΕΠΕ, τέτοια προγράμματα σίγουρα θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο μιας πλήρους ΣΠΕ. Η οδηγία όμως δίνει και περιθώρια ελιγμών τη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη στο άρθρο 3.3 για τη χρήση τοπικών γεών, μικρής κλίμακας γεών. Εκεί μπορεί να μην γίνει πλήρης ΣΠΕ, αλλά μια διαδικασία screening, δηλαδή ταξινόμηση και μια διαδικασία για να αποφασιστεί για το κατά, το πόσο χρειάζεται ΕΠΕ ή ΣΠΕ. Ξεκίνησε λοιπόν και έγινε το screening για το συγκεκριμένο project. Ήταν αρνητικό το συμπέρασμα που αποφάσισαν δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να γίνει πλήρης ΣΠΕ. Αυτή λοιπόν η διακριτική ευχέρεια για το screening αφορούσε και το κατόφλι στην νομοθεσία ΣΠΕ. Δηλαδή 10.000 κάτοικοι είναι το κατόφλι. Χρειάζεται τότε από εκεί και πάνω δηλαδή να υπάρχει ΣΠΕ, αφού δεν ήταν τόσοι κάτι και δεν ήταν λοιπόν ανάγκη. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν μια διαδικασία παραβάσεων όπως σας είπα κατά της Ιρλανδίας για την ε, οδηγία ΣΠΕ. Καταλήξαμε στο ότι ήταν πάρα πολύ ψηλά τα κατόφλια, έχουν αλλάξει τα κατόφλια. Έχουν εισαχθεί επίση αλλαγέ ε, και στην μετάταξη τη οδηγία ΣΠΕ στο δίκαιο της Ιρλανδίας και οι Ιρλανδικέ αρχές ε, δεσμεύτηκαν ότι θα είναι πιο αυστηρές. Εμεί παρακολουθούμε του σύνεγγυ στην υπόθεση. Το θέμα ε, δεν είναι λευκό ή μαύρο ουσιαστικά, ε, δηλαδή αν θα έχουμε μόνο screening ή αν θα απαιτείται πλήρης ΣΠΕ ή ΕΠΕ. Δεν μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι έχουμε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουμε αδιάσυστα επιχειρήματα για να δείξουμε ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση με το screening. Όπως ανέφερα, αυτή τη στιγμή με νέα νομοθεσία ε, δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Πλέον, κατά πάσα το θα γίνονται πλήρης ε, σπέ και δεν θα γίνεται απλά screening. Επίσης, λάβαμε πληροφορίες από τις ε, Ιρλανδικές αρχές σε ό,τι αφορά την ανάλυση κινδύνων. Για τις εγκαταστάσεις έγινε ε, και στο onshore ε, κομμάτι, αλλά και στο πλαίσιο του διασεβέζου. Αυτό που είδαμε όμως ήταν και η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ε, τεκμηρίωση για την ΕΠΕ. Ε, διαπιστώσαμε ότι στην τεκμηρίωση αυτή υπάρχει και μία αξιολόγηση κινδύνων που θα προέρχονται από την μεταφορά υγραερίου μεσοπλίων. Είδαμε ότι υπάρχει λοιπόν και μία ανάλυση θαλάσσιων κινδύνων, κινδύνων και το θαλάσσιο περιβάλλον στο πλαίσιο αυτή τη ΕΠΕ. Βέβαια, δεν έχουμε αναλυτικά στοιχεία για το βαθμό στον οποίο υπάρχουν προβλήματα που αναφέρουν. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι ουσιαστικά επρόκειτο για μία ε, εκτίμηση που δεν είχε καθόλου να κάνει με τους θαλάσσιους κινδύνους, αλλά με, την, ε, ε, με το κατά πόσον μπορούν τα σκάφη να πλέψουν σε αυτά τα ύδατα. Για την πλοημότητα ήταν, δεν ήταν καν για το θαλάσσιο κίνδυνο. Και δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια κριτήρια για τη μεταφορά διαξηράς και τη μεταφορά διαθαλάσσης. Το θέμα είναι ότι δημιουργούμε κάποιες περιοχές επικίνδυνες. Λέμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτή το, την περιοχή, πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό έγινε για την ξηρά, δεν έγινε για τη θάλασσα. Από τη στιγμή που μπορεί να περάσει το πλοίο, δεν σημαίνει ότι είμαστε εντάξει. θα μπορούσε να υπάρχει και μια εγκατάσταση βανθέων υδάτων. Μπορούσε να φτάνει μέχρι το Ρότερνταμ για παράδειγμα, η μεταφορά. και γίνεται λόγος για 500 μέτρα. Δεν μπορεί δηλαδή ξαμενόπλου που μεταφέρει υγραέριο να είναι 500 ε, μέτρα και προς τις δύο ε, πλευρές. Άπαξ όμως και μπουν στον κόλπο, στο, στο δέλτα, ε, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να καλύπτει ενδεχόμενα προβλήματα, ενδεχόμενους κινδύνους. Εγώ είπα να δείτε τον, ε, τη μελέτη για την εξολόγηση των θαλάσσιων επιπτώσεων. Εκπρόσωπος Κομισιόν, ναι, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Obviously, ε, they are... Όπως καταλαβαίνετε, ναι, πράγματι υπάρχουν στοιχεία ε, στη θαλάσσια, στην εκτίμηση θαλάσσιου κινδύνου. Όχι ότι δεν έχει τίποτα αυτή η ΕΠΕ, το θέμα είναι κατά πόσον εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε του διαφορετικού αυτοθερματικού σταθμού υγραερίου και να εξετάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο εξολογήθηκαν οι κίνδυνοι για το θαλασσιο περιβάλλον ή να δούμε σε ποιο βαθμό αν συγκρίνουμε την τεκμηρίωση από την ευαλική περίπτωση με την ελληνική περίπτωση, να δούμε αν είναι ζήτημα βέλτιστης πρακτικής των αρχών που σχεδίασαν, που μελέτησαν και των αρχών που εκτελούν. με βάση την αναφορά, την ανακοίνωση μάλλον για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, την ανακοίνωση μας για την αναφορά από το Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω ότι υπάρχουν τώρα χάρτες, καταρτίζονται ειδικοί χάρτες. Και τώρα αυτό αν μπορεί να επιβληθεί στο Σάνον για την περίπτωση εκεί του Δέλτα ή αν αυτό υπερβαίνει τις απαιτήσει της οδηγίας ΕΠΕ ή αν εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε. Ε, Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε αναλυτικά τα επιχειρήματά σας και τα αναλυτικά έγγραφα. Σας ευχαριστώ που το πάρω. Εκτός μικροφώνου. Uh, thanks very much and thanks to the petitioner and to the, the commission. Ευχαριστώ πολύ και τον αναφέροντα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι αυτή η αναφορά αποτελεί προηγούμενο συνήθες στην Ιρλανδία, δυστυχώς, όπου υπάρχουν πολλά project που διευθύνονται από μεγάλους οργανισμούς, οργανισμούς φυσικού αερίου και υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι απομονωμένες, ακατοίκητες όμως και οι λίγοι κάτοικοι που έχουν αυτές οι περιοχές θα έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Οι κάτοικοι αυτοί αγνοούνται από αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς που ε, εκτελούν αυτά τα project και η κυβέρνηση δυστυχώς ακολουθεί και το ίδιο σκεπτικό. Σύμφωνα με την Επιτροπή ότι υπάρχει η ανάγκη για στρατηγική ΕΠΕ, για ΣΠΕ, αλλά μου φαίνεται δύσκολο και μου φαίνεται κάπως περίεργο επίσης το ότι οι άνθρωποι που μένουν στις λιγότερο κατοικημένες περιοχές, αεροκατοικημένες, να έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους άλλους. Έγινε και μία παρόμοια περίπτωση στην Δυτική Ιρλανδία, σε μία αεροκατοικημένη περιοχή, όπου αγνοήθηκαν παντελώς οι ανησυχίες του, των κατοίκων εκεί και η εφαρμογή της σχετικής οδηγίας. Μου φαίνεται πως από αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορώ να εξάγω τα εξή. Εάν αυτό δεν μπορεί να συμβεί από εδώ και στο εξή, δεδομένης της αλλαγής της νομοθεσίας στις, ε, στην Ιρλανδία και θα υπάρχει λοιπόν ε, υποχρεωτική ανάγκη για διεξαγωγή ΣΠΕ, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και δεν θα υπάρχει επομένως λόγος να υποφέρει, να υποφέρουν οι κάτοικοι της κοινότητας αυτής από τις αρνητικές επιπτώσεις, διότι έχουν δικαίωμα για διεξαγωγή. Επίσης, ο αναφέρον σαφές ότι, καθιστά σαφές ότι η διεξαγωγή ε, εκτίμηση θαλάσσιου κινδύνου είναι ανεπαρκή. Η κατασκευή του έργου αυτού έχει τεράστιε επιπτώσει όχι μόνο στην ξηρά αλλά και στη θάλασσα και χρειάζεται να γίνει σωστή εκτίμηση του κινδύνου. Φυσικά και θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, αλλά εγώ θα πρότεινα να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να συνεργαστούμε, να κάνουμε επίσκεψη στην Ιρλανδία. Νομίζω θα γίνει τον επόμενο Σεπτέμβρη και τότε θα είναι μια καλή ευκαιρία για, τα, για τους ευρωβουλευτές να δουν την κατάσταση και να μιλήσουν και με αυτούς που τους αφορά το θέμα στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Um, thank you very much. Would you like to add something? Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Κύριε Μποστινάρου. Σήμερα το πρωί, βλέπετε, συζητούσαμε όλες τις τροπολογίες για, την, για τις ΕΠΕ. Και τουλάχιστον τώρα, με αυτές τις ε, τρεις περιπτώσεις, αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να τροποποιηθεί η οδηγία για τις ε, ΕΠΕ, έτσι ώστε να αποφύγουμε προβλήματα όπως αυτό που συζητούμε τώρα. Ας δούμε τώρα το περιεχόμενο της αναφοράς. Υπάρχει προηγούμενο. Το Milford Haven. Και εάν ήταν καλό προηγούμενο τότε, γιατί δεν είναι καλό προηγούμενο τώρα στην περίπτωση του Σάνων. Γιατί μας το λέτε αυτό. Αυτό τι δείχνει ότι η ΣΠΕ με τον τρόπο που διεξάγεται τώρα, δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί ερωτηματικά. Τι γίνεται, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καλό, σε ορισμένες περιπτώσεις όχι. Γιατί δεν μπορούμε να το εφαρμόζουμε σε κάθε παρόμοια περίπτωση με αυτή του Milford Haven. Μετά, δεύτερον. Σίγουρα η φορά πρέπει να μείνει ανοιχτή. Εγώ θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί σκληρότερα διότι βλέποντας ε, το περιεχόμενο της αναφοράς φαίνεται ότι οι επένδυτες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν έχω πρόβλημα με τους επενδυτές ε, από, τα, από τις νήσους ε, Καϊμάν. Έχω όμως πρόβλημα με, το, με τα γεγονότα, διότι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν πραγματικό υπόλογο, ότι η λογοδοσία θα ισχύσει. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι εάν ε, συμβεί κάποια φυσική καταστροφή, κάποιος θα καλύψει το οικονομικό κόστος και όχι μόνο. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τόσο προηγμένοι όσον αφορά τους φορολογικούς παραδείσους, αλλά τι θα γίνει εάν μετά από ένα-δύο χρόνια εξαφανιστούν αυτοί οι επενδυτές και το μόνο που μένει από αυτούς είναι μια ταχυδρομική θηρίδα που δεν θα απαντά σε καμία επιστολή από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι θα γίνει τότε. Αυτό είναι το σύνηθε. Έτσι λοιπόν, η λογοδοσία, οι οικονομικές εγγύησεις πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, διότι θα γίνουν οι καταστροφές, θα υπάρχουν ζημιές σε μεγάλη κλίμακα και σε περίπτωση που συμβεί αυτό κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτός που μολύνει πληρώνει. Αυτή είναι η αρχή. Και στη δική μου έκθεση για τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής προτείνω να ενισχυθεί το ότι ο Μολύνων πληρώνει. Και προτείνω να μην υπάρχει η δυνατότητα να καλύπτεται το κόστος παρομοιών περιπτώσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να συνάδει με αυτό, με το ότι ο Μολύνων πληρώνει και να εγγυηθεί και να φροντίσει ώστε το οικονομικό υπόλογο θα επιληθεί. Διότι δεν ξέρω, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είμαι και τόσο σίγουρος και τόσο αισιόδοξο. Σας παρακαλώ, έχει... θυμηθείτε, δεν είμαστε κόλπος του Μεξικού και Ηνωμένε Πολιτείε εναντίον της British Petroleum. Ξέρετε πόσα χρήματα αναγκάστηκαν να πληρώσουν για αποζημιώσεις. Ποιος θα πληρώσει σε παρόμοια περίπτωση, άμα γίνει κάτι εδώ. Και όχι μόνο αυτό, είναι υποχρέωση όχι μόνο του κράτους μέλους, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που εγγυείται την σωστή εφαρμογή των συνθήκων και πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτό θα γίνεται μόνιμα και συνεχώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ποστινάρου. Ήταν πολύ σοφή η ολοκλήρωση της συζήτησης. Έχω να προτείνω κάτι και στους δύο σας, διότι είστε οι μόνοι οι ευρωβουλευτές που βρίσκονται εδώ τώρα από αυτή την Επιτροπή. Έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές αναφορές, όπως αυτές που κοιτάξαμε σήμερα το πρωί. Αυτές οι αναφορές προτείνω να σταθούν στην Επιτροπή ΕΝΒΙ, διότι έτσι, ενδεχομένω, η Επιτροπή Ένβη να μπορέσει να βρει τα διάφορα νομικά κενά. Συμφωνείτε, κύριο Γιάρ. Συμφωνώ απόλυτα με την προϋπόθεση να προσέξουμε να λάβουμε απάντηση εν ευθέτω χρόνο. Όχι κάποτε. Πολύ με ενδιαφέρει η γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής αυτής, αλλά όχι σε ένα χρόνο σύντομα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω οι πρόεδροι των Επιτροπών να βρίσκονται σε επαφή. Ευχαριστώ. I Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τους διερμηνείς και τους αναφέροντες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα σας.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 και βεβαίως μετά θα το αφήσουμε ανοιχτό σε εσά για να δούμε τι ε, θα κάνετε όταν θα έχετε και όλη την ε, ανεργική γραπτή μας έκθεση. Βεβαίως, αν υπάρχουν ε, περαιτέρω ζητήματα, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, ως Ελληνίδα, εγώ αισθάνομαι λίγο αμήχανη, αλλά παρόλα αυτά ε, νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές έτσι ώστε να ζητήσουμε τελικές απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Um, just from the B part to the A Σχετικά ε, με την 23, 26, 51, 59 θα θέλαμε να τις κρατήσουμε ανοιχτές. Ε, επομένως να μην τις βγάλουμε από τον κατάλογο που έχουμε εδώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.